Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Εννιά και 4 λεπτά να ξεκινήσουμε. Άρχεται λοιπόν η συνεδρία της Επιτροπής μας και να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης η μακροοικονομική υποστήριξη που πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία. Είμαστε σε δεύτερη φάση εξέτασης του θέματος και έχουμε ένα νέο κείμενο. Ο εισηγητής μας κύριος Λαντσμπέργκης μας υπέβαλε τον νέο κείμενο Έχουμε εντωμεταξύ 43 τροπολογίες και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο στάσεις έναντι του, έναντι του θέματος αυτού ορισμένοι που θα πούν ότι είναι πολλά 1,8 δις για την Ουκρανία, ότι θα μπορούσαμε να τα δαπανίσουμε με καλύτερο τρόπο και άλλοι θα πούν ότι δεν αρκούν, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Εγώ βεβαίως ε, πιστεύω ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, καλύτερα, ταχύτερα. αλλά σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας το θέμα ήταν ε, να τους χορηγήσουμε το ταχύτερο δυνατό βοήθεια. Να βοηθήσουμε μια χώρα που προσπαθεί να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις ενώ είναι σε πόλεμο για να διαφυλάξει την εδαφική της ακαιρεότητα. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, από τις πολιτικές ομάδες, ε, από όλες τις τάσεις που ε, μας βοήθησαν να έχουμε αυτήν την ταχεία χορήγηση βοήθειας και που συμφωνούν ότι πρέπει να εγκριθεί αυτή η βοήθεια όσο το δυνατόν ταχύτερα ή δυνατόν ε, να αποσταλεί ήδη το καλοκαίρι. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους της ΑΦΕΤ που ενέκριναν την γνωμοδότηση της Επιτροπής τους η οποία γνωμοδότηση και αυτή συμφωνεί με αυτό το βασικό θέμα της ταχείας διαδικασίας. Και αυτό θα είναι και το ισχυρότερο μήνυμα. Δεν θα είναι ότι είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που έδωσε ποτέ η Ένωση σε τρίτη χώρα. Το ισχυρότερο μήνυμα θα είναι ότι η Ένωση, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε όλοι επ' αυτού, αλλά στην τελευταία συζήτηση εγώ αυτό απεκόμισα τουλάχιστον, ότι ήμασταν ενωμένοι. Δεν ακούσαμε απόψεις που, ήταν, που θα ήσαν κατηγορηματικά κατά της ε, αποστολής βοήθειας στην Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε περήφανοι για αυτό το μήνυμα και αυτό το μήνυμα να δώσουμε και στους φίλους μας στην Ουκρανία ότι ήμασταν και θα είμαστε ενωμένοι. Να ψηφίσουμε λοιπόν με το ίδιο πνεύμα που ψηφίσαμε που συζητήσαμε και κατά την προηγούμενη συζήτηση και σας ευχαριστώ για αυτή την θαυμάσια δυνατότητα. Αυτά ευχαριστώ. Ας περάσουμε αργότερα στην ψηφοφορία. Πρόεδρος. Από τους Σκιώδης, ο Μποστινάρου δεν είναι παρόν, ο κύριος Πίχα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λαντσμπέργκης για την σωστή διαδικασία για αυτό το θέμα που είναι τόσο καυτό και επίκαιρο. Είπαμε στη, στην Πολωνία έχουμε μια έκφραση που λέει ότι η ταχεία βοήθεια είναι διπλής αξίας. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Είναι τραγική κατάσταση της χώρας. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε σύντομα. Ευχαριστώ την Κομισιόν επίσης που υπέβαλε το έγγραφο αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ε, πραγματικά με καλό τρόπο την Ουκρανία διότι προτείνει ψηλό ποσό βοήθειας και περιγράφει και τους όρους ε, παροχής αυτής της βοήθειας. Η ομάδα μου, το ECR, υποστηρίζει συνολικά την πρόταση. Πρέπει να δοθεί η βοήθεια και φυσικά επιγόντως, ταχύτατα. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Λαντσμπέριξ, αλλά να προσθέσω ότι όχι απλώς αγωνίζονται για την εδαφική τους ακαιρεότητα, αλλά και για την κυριαρχία τους. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Φανμπάλεν. Α, εσείς θα τον εκπροσωπήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας συμφωνεί με τον εισηγητή. Πρέπει να αποφασίσουμε ταχύτατα Οπότε, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των πολιτικών ομάδων, δεν θα υποστηρίξουμε καμία τροπολογία και ε, να σα θυμίσω ότι συμφωνεί και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Χαλμούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα είμαι σύντομο. Αλλά όχι τόσο σύντομο, όσο οι προηγούμενοι. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε αν η άποψη μέχρι τώρα του Κοινοβουλίου χωρίς να ελέγξει τι γίνεται να αποφασίζει για τα θέματα της Ουκρανίας και να δίνει αυτή τη βοήθεια, αν είναι η καλύτερη. Νομίζω Ω Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, που έχει λοιπόν ε, εξωτερικέ αρμοδιότητε, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την κατάσταση στην κοινωνία τη ε, στην Ουκρανία να δούμε και τις πολύ περίπλοκες σχέσεις μεταξύ ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας Ουκρανίας Ένωσης και άλλων ε, σημαντικών παραγόντων της διεθνούς πολιτικής. Γιατί δεν είναι μόνο ένα, ένα γενικό θέμα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της Ουκρανίας. Το θέμα είναι με τι τρόπο και κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, απαιτήσει να υπάρχει και αιρεσιμότητα. Θέλω να τονίσω ότι και εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι μια λειτουργική δημοκρατική χώρα με τις κατάλληλες δομές και να μην επηρεάζονται οι κοινωνικές δομές και η εξουσία από την επιρροή των ολιγαρχών και να μπορούν όλοι οι πολίτες ε, κυρίαρχα να αποφασίζουν για τη χώρα τους σε μια χώρα με πλήρη κυριαρχία. Και κατά τη διαδικασία που έχουμε τώρα, λόγω του τρόπου με τον οποίο έγιναν οι συζητήσεις για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης, φέρει ευθύνη και η Ένωση. Τρία συγκεκριμένα θέματα της ε, έκθεσης Λατσμπέργης θέλω να συζητήσω. Πρώτον, η πρόταση της Κομισιόν αναπτύσσει την αιρεσιμότητα με κριτήρια που έχουν αποτύχει στο εσωτερικό της Ένωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεύτερον, οι αμφιβολίες μου λοιπόν είναι εάν θα πρέπει να δώσουμε 1,8 δις στην Ουκρανία ως δάνειο σε αυτή την φάση εφόσον ε, συζητάμε και ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο θα συμπεριλαμβανόταν και αυτή η βοήθεια. Είναι ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 15 δις. από ό,τι φαίνεται οι ανάγκε της χώρα είναι γύρω στα 40 δις. Αλλά δεν είναι αυτή μόνο η ουσία του προβλήματο ήδη αναφέρθηκε. Όπω λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ουκρανία ποτέ δεν θα μπορέσει να επιστρέψει αυτό το δάνειο. Άρα θεωρούμε όλοι ότι κατόπιν θα γίνει κάποιο κούρεμα του χρέους. Εφόσον αυτή είναι η συνολική εικόνα, Τότε τίθεται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα, τι θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον. Δηλαδή θα δίνουμε χωρίς να συζητάμε και χωρίς να θέτουμε προϋποθέσεις διάφορα ποσά, γνωρίζοντας ότι ε, στην ουσία είναι η ίδια λογική με αυτήν την οποία υιοθετήσαμε για την Ελλάδα. Δηλαδή ότι δίνουμε ποσά επειδή υπάρχει πήγουσα βοήθεια χωρίς να ξέρουμε αν μπορούν να επιστραφούν. Στην ε, ε, πρόταση της Κομισιόν το δάνειο αυτό συνδυάζεται με αίτημα για να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Όμως η ηγεσία της Ουκρανίας πάντα ανακοινώνει επιτυχίες στην καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Όμως στον προϋπολογισμό της ε, Ουκρανίας για το 2015 δεν λέγεται τίποτα για τη δημιουργία μιας αρχής κατά της διαφθοράς και από ό,τι ξέρω σταμάτησε η διαδικασία πρόσληψη υπαλλήλων προς αυτή την κατεύθυνση με οδηγία από τα ανώτατα κλιμάκια. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει με την Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας μας υπέβαλε ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε με πάρα πολλά μέτρα. Όμως λόγω της ε, σύγκρουσης στον Τόνμπας καταλαβαίνουμε την κατάσταση θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας Μίνσκ 2. Αλλά θεωρούμε ότι ερμηνεύουν διαφορετικά οι αρχές της Ουκρανίας αυτή την, ε, την συμφωνία. Είναι ένα θέμα εσωτερικού σχετισμού δυνάμεων στην Ουκρανία. Δύο παραδείγματα. Μετά τις συζητήσεις του Προέδρου με την Γερμανίδα καγκελάριο υπόθηκε από τον κύριο Ποροσέγκο ότι απέτυχε η συμφωνία Μίνσκ 2. Αλλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Δεύτερο παράδειγμα. Οι ομάδες των εθελοντών έχουν ε, διαφοροποιηθεί από την ε, συμφωνία Μίνσκ 2 και θέλουν να είναι αυτοί οι μόνοι οι οποίοι διεξάγουν αυτή τη μάχη. Αυτή η εθνοφρουρά όμως αυτή τη στιγμή δαπανούν το μεγαλύτερο τμήμα του αμυντικού προπολογισμού. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ε, πώς ακριβώς θα βοηθήσει αυτή η οικονομική βοήθεια. Είναι λοιπόν πολύ περιπλοκή, πολύ πιο περιπλοκή η κατάσταση από ό,τι έχει περιγραφεί μέχρι τώρα και γι' αυτό υπέβαλα τροπολογία που θέλει να δημιουργήσει μια σαφή αιρεσιμότητα Δηλαδή να μην αξιοποιηθούν αυτά τα ποσά για μη ειρηνικού σκοπούς. Ξέρω τη θέση των άλλων πολιτικών ομάδων και των συναδέλφων στην Επιτροπή. Λυπάμαι που δεν συζητάμε σοβαρά αυτό το θέμα και θεωρώ ότι είναι αυτό σοβαρό πολιτικό σφάλμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Βίκτορ Μποσινάρο, τώρα έχει το λόγο, γιατί έχει καταστάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας και να πω ότι οι σοσιαλιστές θα υποστηρίξουν ε, την πρόταση Λαντσπέργκης χωρίς τροπολογίες. Μόνο και μόνο για να διασφαλίσουμε ότι θα ε, εγκριθεί με την ταχεία διαδικασία η έκθεση Κατά δεύτερον, είναι εξίσου σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να εγκρίνουμε την έκθεση έχοντα υπόψη και τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ουκρανία και την κατάσταση που επικρατεί στην ε, Ουκρανία κατά τρίτον. Εξίσου σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί το πλέον ενδεγμένο κλίμα και την πλέον ενδεγμένη ατμόσφαιρα να εφαρμοστεί πλήρως σε μια συμφωνία ούτε στην Ουκρανία ούτε σε καμία άλλη χώρα. Αλλά εγώ παρακαλώ τους αγαπητούς συναδέλφους που ανέφεραν τον πόλεμο είναι να σκεφτούν ποιος ξεκίνησε, επέβαλε τον πόλεμο, ποιος πήρε κομμάτια της επικράτειας της Ουκρανίας που αναγνωρίζονται το διεθνές δίκαιο. Και τέλος να σημειώσουμε το εξή. Σε καιρό πολέμου για την Ουκρανία και ενώ πολλοί δυτικοί εταίροι της Ουκρανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ, ΕΕ, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιο πολλά εν περιπτώσει, προσπαθούν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Σημειώνουμε ποια μέτρα έχει λάβει η Ουκρανική κυβέρνηση και είμαστε και σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας αναφέρουν όλες οι υπηρεσίες αυτές μεγάλο αριθμό, μεγάλη σειρά άλλων ε, ειδικών που ε, συνδράμουν την Ουκρανική κυβέρνηση για τις καλές πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν από την Ουκρανική κυβέρνηση είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό επίπεδο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλες αυτές τις πτυχές ε, από πλευράς της ομάδας μου σας δηλώνω ότι θα υποστηρίξουμε την έκθεση του κ. Λανσπέργκης. Δεν θα καταθέσουμε τροπολογία, συμφωνούμε με την ιδέα αυτή και θα υπερψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή στο τέλος, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε αλληλεγγύη με μια χώρα, με ένα έθνος, σε καιρό πολέμου, πολέμου από τον οποίο ξεκίνησαν άλλοι και όχι οι Ουκρανοί. Ε, pour le groupe des Verts, ε, για ε, τους πρασίνους. Θα υποστηρίξουμε την ε, επιταχυμένη διαδικασία. Αν και για μας ε, είναι όλο και πιο ζώρικη η κατάσταση. Διότι υπενθυμίσαν ορισμένοι ότι βεβαίως λόγω της κατάστασης είναι βασικό καθήκον για την Ένωση να στηρίξει την Ουκρανία και οι πιέσεις ο πόλεμος που λαμβάνει η χώρα εκεί μας υποχρεώνει να δράσουμε ταχαίως. Ωστόσο, σε κάποια φάση θα πρέπει να εξετάσουμε και το Κοινοβούλιο συνολικά να εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Γιατί δεν έχουμε ακόμη όλες τις δυνατότητες να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η καλύτερη βοήθεια για να δώσουμε στην Ουκρανία. Ο Χέλμουντ το υπενθύμησε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ουκρανικό χρέος. Συνεχίζουμε να τους δίνουμε δάνεια. Οι δυνατότητες ε, βοήθειας μέσω των μέσων γειτονίας ε, δεν αξιοποιούνται ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θέτουμε αρκετές προϋποθέσεις. που θα μπορούσαμε παρά την ιδιαίτερα δυσχερή για τις αρχές κατάσταση να τις θέσουμε. Όλο και περισσότερο λοιπόν ε, περιπλέκεται η κατάσταση. Γιατί ναι, λέμε πρέπει να αντιδράσουμε ταχαίως, ναι, να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά αποτελεσματική κατά το δυνατόν. Και δεν ε, πιστεύω ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να αποφασίσουν κυρίαρχα και δημοκρατικά παρά τον πόλεμο που ενορχιστρώνει η Ρωσία. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση, ταχεία αντίδραση, αλλά για μας, για να σας πω την αλήθεια, είναι όλο και πιο δύσκολο για μας να βοηθήσουμε ε, με βάση μια προσέγγιση που δεν μας επιτρέπει να επέμβουμε επί της ουσίας. Ο κύριος Σοπάτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφε, βρίσκεται σε κάποιον πάρα πολύ σοβαρό εμφύλιο πόλεμο η χώρα αυτή και ο λόγο είναι η άρνηση των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν υπόψη την ιστορική τη ταυτότητα, αλλά και τι γεωπολιτικέ διαστάσει τη χώρα αυτή που είναι μεταξύ Δύση και Ανατολή. Προ τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να τραβήξουμε και γι' αυτό εξωθήσαμε την ε, Ρωσία να αναλάβει την υπεράσπιση του πληθυσμού που στην ε, Ανατολική Ρωσία. Ρωσία νεκρή, η οικονομία διαλυμένη και έχουμε μια ύφεση 7% το 2014, τώρα έχουμε ένα έλλειμμα τεράστιο του 12% και επίσης να δούμε τι έγινε και με, το, με την Εύτο και έχουμε αυτή την αυτοκτονική κυβέρνηση του Κιέβου το οποίο έχει κλείσει τη στρόφιγγα για όλες τις παραχές προς τους πολιτισμούς αυτούς του, της Ανατολής και έτσι τα πράγματα τα παραξύνει. Να, ποια, είναι ο απολογισμός των έχουμε κάνει, τι, έχει κάνει, τι έχουν κάνει οι Βρυξέλλες και η Washington και οπότε όλοι, όλα αυτά τώρα θέλουμε να ρίξουμε χρήμα, περίπου ένα δις το 2015 και μιλούμε για σταθερότητα, για ανάπτυξη, να σαν να μιλάγαμε για την Ελλάδα. Μιλάμε για μια χώρα μέσα σε χάο γεωπολιτικό και μιλάμε για μια χώρα που ένα σκοτώνει τον άλλο. Οπότε το θέμα δεν είναι το χρήμα. Δεν θα φέρει αυτό την ειρήνη στη χώρα. Γιατί το να ρίξουμε χρήμα σε μια χώρα που κατάσταση είναι εμπόλεμη είναι σαν να θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε περισσότερη εμπόλεμη κατάσταση. Χρειάζεται μια συμφωνία θα πρέπει να σταματάμε να περιφρονούμε έναν τόσο σημαντικό παράγοντα διεθνή όπως τη Ρωσία και αυτά τα χρήματα, κύριε Λαντσμπέργκης, δεν θα ωφελήσουν, δεν θα σπρώξουν τη χώρα προς ανάπτυξη και σταθερότητα. Πρόκειται να πάνε για αγορά όπλων, ούτω ώστε να υπάρχει ένας στρατός καταστολής, όπως ξέρετε, ένα στρατό που βομβαρδίζει το λαό. Κυρίε και κύριοι, πρόκειται για αυτού οι οποίοι δίνουν τη μάχη τους αυτού που του ονομάζεται επαναστάτε για να προστατεύσουν το χωριό του, τα παιδιά του αλλά είναι πολύ πιο αποφασιστική από τον Ουκρανικό στρατό που βρίσκονται μακριά από το, το, το, το, το δικό του τόπο καταγωγή και δεν έχουν το δίκαιο με το μέρο του. Επομένω, αυτό που χρειάζεται είναι όχι να πλουτίσουμε κάποιου, αλλά χρειάζεται να κάνουμε κάτι για την ε, ειρήνη. Όχι να ενισχύσουμε κάποιου παράγοντε του Κιέβου, όπω προχωρούν τη χώρα στον Κρεμό. Äh, äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να διευκρινίσω από πλευρά τη ομάδα μα το εξή, ότι ε, αποστασιοποιούμεθα από τι δηλώσει του προηγούμενου μιλητή και του κυρίου Σόλτ. Γιατί οι υπεύθυνοι για τα προβλήματα, όχι για όλα τα προβλήματα, γιατί τα πιο πολλά όμω προβλήματα τη Ουκρανία σήμερα είναι η κατοχή ε, τμήματων της χώρας είναι άλλοι ε, παράγοντες και νομίζω ότι εκπρόσωποι ενός, μιας ομάδας που χρηματοδοτείται από ρωσικές ε, τράπεζες δεν θα έπρεπε να παίρνουν το λόγο και να μιλούν εδώ. Äh, Ο Πρόεδρος, να δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κ. Στεμπράνο. Hm. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τη θέση του εισηγητή να προχωρήσουμε γρήγορα και να περάσουμε στην έγκριση της ε, πρότασης αυτής χωρίς τροπολογίες, το οποίο και υποστηρίζουν οι πιο πολλοί σκιώδεις και όπως ανέφερα και στο παρελθόν η κατάσταση μακροοικονομικής χρηματοπιστικής κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει κρίσιμη και στο πλαίσιο αυτό όπως ξέρετε η Διεθνής Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα πρόγραμμα ε, χρηματοπιστωτικής βοήθειας για 17 δισεκατομμύρια και τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω παρά την προηγούμενη σταθεροποίηση αλλά και τα επιτόκια αποτυπώνουν την κρίση αυτή και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα του Διεθνού ε, Νομισματικού Ταμείου και θεωρούμε λοιπόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα για την εφαρμογή τη αρρωγή αυτή. Για τα σχόλια του κυρίου Σόλτ, θα ήθελα να σχολιάσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λαμβάνει υπόψη ασφαλώ ε, τα σχόλια αυτά και τις ανησυχίες του και θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το Κοινοβούλιο ότι σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα στα πλαίσια του προγράμματος αυτό. Ε, κοιτάμε την πολιτική κατάσταση και είμαστε κοινωνικά, δείχνουμε κοινωνική ευαισθησία. Να τονίσουμε την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ε, βοήθειας και επίσης συνυπολογίζουμε πάρα πολύ την ενίσχυση της, των δημοσιονομικών της Ουκρανίας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο εισηγητής έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Για να απαντήσω στα σχόλια, πρώτα-πρώτα, για τον κύριο Σόλτσο τα επιχειρήματά σας τα έχω ξανακούσει σε σχέση με το πού θα πρέπει να κατευθύνουμε τα χρήματα. Γιατί εάν το timing ήταν σωστό, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό όσο χρειάζεται. Εγώ θα ήμουν ο πρώτο που θα έκανε αυτή την κουβέντα. Γιατί νομίζω ότι είναι λογικό και στέκει. Όμω το θέμα τώρα είναι ότι η χώρα δίνει τη μάχη για την ύπαρξή τη, την ακυρότητά τη. Και έχουμε δύο ηγέτε τη Ένωση που πήγαν στο Μίνσκ και είπαν Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για να σταματήσει ο κόσμος να σκοτώνεται και να σταματήσουν να καταστρέφονται οι πόλεις. Να τι χρειάζεται τώρα. Αυτό ελπίζουμε. Αν μπορούμε να το πετύχουμε, τότε μπορεί να αρχίσουν και οι μεταρρυθμίσει. Ενθαρρυντικά ήταν αυτά που διάβασα. Ότι στη Ράντα πέρασαν οι μεταρρυθμίσει. Και αρχίζει η υλοποίηση αυτών. Επομένως, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε το πώς και πού θα δώσουμε την υποστήριξή μας, αν θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα, λιγότερα, να υποπτεύσουμε ή όχι. Χρειάζεται επομένω σταθερότητα, να σταματήσουν οι άνθρωποι να σκοτώνονται. Τώρα, ακούμε συνέχεια το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φταίει για τα όσα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτό άπαξ και δεπαντός να σταματήσει γιατί δεν υπάρχει στρατός της Ένωσης ή στην Ουκρανία. Δεν καταλάβαμε εμείς την Κρυμαία. Δεν ήμασταν εκεί όταν αυτά γίνανε. Άλλοι τα έκαναν αυτά. Άρα να, σταματάμε, να σταματήσουμε αυτή την αυτοκατηγορία. Εμείς είμαστε εκείνοι που βοηθούν και να είμαστε υπερήφανοι. Σας ευχαριστώ και θα ψηφίσουμε στις 10 για το θέμα αυτό. Και περνάμε λοιπόν στο σημείο 9 της σημερινής έταξης. Το θέμα της των ε, χωρών της, των Δυτικών ε, Βαλκανίων, της Βοσνίας Αρζεγοβίνης ιδιαίτερως ε, και των εκ των εμπορικών μέτρων. Έχουμε σχετική έκθεση. Επτά τροπολογίες κρατέθηκαν. Τέσσερις από τη γνωμοτότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τους Συναδέλφου για τη συνεργασία του όσον αφορά την έκθεσή μου και ευχαριστίε ακόμη περισσότερε στον συνάδελφο Στήρ που ήταν ο όλοι συζητητή για την ευφυή e του βοήθεια, τι ικανότητε του και για το πόσο ήταν διαθέσιμο για να συνεργαστούμε. Όπω γνωρίζετε, πρόκειται για μια έκθεση που έχει να κάνει με πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μια τροποποίηση κανονισμού του 2009 που αφορά τη σταθεροποίηση των μονομερών προτιμήσεων εμπορικών όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Και προτείνονται εδώ κάποιες τροποποίησεις ε, βασικά, βασικά σημεία είναι οι, οι εμπορικέ προτιμήσει αυτέ να επεκταθούν και προ αυτέ τι χώρε μέχρι το 2020. Επίση υπάρχει κάποια σημαντική ρήτρα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτείνει αναστολή για Βοσνία και Ερζεγοβίνη από 1η Πρώτου του 2016 αυτή τη συμφωνία που προτείνωσαν εάν δεν εγκριθεί η ενδιάμεση συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν της ε, προσχώρησης της ε, Κροατίας. Όπως έχουμε πει το πρώτο θέμα εδώ είναι το ότι στην έκθεση επαναλαμβάνουμε το ότι αυτή η πρόταση της Προεδρικής Επιτροπής για αναστολή της Συμφωνίας Προτιμήσεων είναι κάτι το θεμητό. Και επίσης αποτυπώνει πώς είναι το τοπίο Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις. Τι ίσχυε πριν την προσχώρηση της Κροατίας. Επομένως δεν υπάρχει εδώ κάποια διαφορά για την Βοσνία. Υπάρχουν παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και Επομένω, δεν υπάρχει κάποια διαφορά τώρα που προσχώρησε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω, υπέστη κάποια ζημία η Κροατία από τότε που προσχώρησε γιατί έχει υποστεί κάποιες επιβαρύνσεις και ήταν η συνέπεια του ότι έπρεπε να πετύχει τους ευρωπαϊκούς της στόχους. Άλλο τώρα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ανθρώπινη την Ευρωπαϊκή Τροπή είναι σύνομα και θα πρέπει επομένω να δούμε με κάποιο είδου τροπολογίες πώς θα ρυθμίσουμε την προοπτική της προσχώρησης της Βοσνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, Γιατί η Βοσνία είναι χώρα στρατηγικής σημασίας. Έχει κάποια ιστορία και μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει, δεν μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο. Επομένως αυτό που χρειάζεται είναι ε, κάποιο είδους παραπάνω πολιτική βοήθεια για να σπροχθεί η χώρα προς αυτή την τόσο σημαντική κατεύθυνση. Και κατά την εκπόνηση της έκθεσης εμείς πασχίσαμε να βοηθήσουμε στα όσα έκανε η Επιτροπή στην Βοσνία, στα όσα έκανε η κυρία Μογερίνη, η πατή και εγκρίναμε ε, την έκθεση για την ε, αξιολόγηση της πορείας της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα δεν είναι να αναλάβει κάποιο τιτάνιο ε, έργο η Βοσνία, αλλά να αναλάβει και να πετύχει κάποια πράγματα εφικτά. Έχουμε επίσης ε, κάποιο έγγραφο, το προσυπέγραψαν όλοι οι ηγέτες της χώρας, το ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας και επομένως αυτό αποτελεί δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις. Και έτσι το Συμβούλιο βρέθηκε σε θέση να δώσει το πράσινο φως όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή και Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικό αυτό. Στο εγγραφό εκείνο, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, ταυτόχρονα καλείται η χώρα να προσαρμόσει τις εμπορικές της σχέσεις. αυτά το οποία τώρα θέλουμε κι εμείς. Άρα αυτοί αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες, αυτοί είναι οι στόχοι των βασικών τροπολογιών. Αυτά τα συζητήσαμε όλες οι πολιτικές ομάδες νομίζω αρκετά ανοιχτά και σοβαρά. Όπως σας είπα, έχουμε τις προπολογίες σε σχέση με μια αξιολόγηση της ε, πολιτικής πορείας της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και τις σχετικές τροπολογίες. Και, κατά δεύτερο λόγο, Έχουμε τις υ πράξεις. Έχουμε κάποιες παραμέτρους στην ε, υπόθεση αυτή. Γιατί εδώ σε κάποια θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει σημαντικά περιθώρια ενέργεια στην ε, χώρα. Οπότε και το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει τον έλεγχό του. Επίσης, εμείς προτείναμε ένα συμβιβασμό. Πρόκειται για τροπολογία του Στίερ. Στην τροπολογία αυτή τονίζει ότι χρειάζεται να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τη χώρα. Ιταλός είμαι και τα έχουμε πει και εμείς στη χώρα μας το μήνυμα που κάνουμε τα ίδια. Οπότε είπαμε για αυτή τη συμμαστική τροπολογία, αυτό το συμβασμό που πρέπει να γίνει αποδεκτός. Ότι δηλαδή τι, θα γίνει τέλο πάντων με, με, με, με τη συμβολή της ε, Βοσνίας σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις πριν προσχωρήσει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά έχουμε την τροπολογία των ανθρώπινων δικαιώματων που συζητήθηκε πολύ και εδώ καλύψαμε ε, καλά, το, την αποσύρω, την αποσύρω όμω. Γιατί στην αρχή το θέμα ήταν κατά πόσον πρόκειται να αντιστραφεί αυτό το επιχείρημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή να μην είναι αρνητική διατύπωση, αλλά θετική. Και κάπω ε, να είναι πιο, πιο δόκιμη η διατύπωση. Ε, μην έχουμε επανάληψη, μην έχουμε επιθετική διατύπωση σε σχέση και με τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πάντω, εγώ αποσύρω την τροπολογία αυτή, γιατί νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε τελικά. Πώς. Έτσι με αυτή την ρήτρα ανθρωπινών δικαιωμάτων θα ήταν δυσκολότερη η υλοποίηση των κατεξοδότηση πράξεων γιατί θα είχαμε διαπιστώσεις διαφόρων ούτως υπήν παραδιάσεων που θα αποσταθεροποιούσαν το κλίμα Πάντως, με την πολύτιμη συνεργασία του κ. Στήρη είπαμε να το αποσύρουμε αυτό και να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και το, κείμενο των πράσινων, του Μπούχνερ, ο οποίος και εκείνος συνέβαλε στη σύνταξη της έκθεσης για μεγάλη υπομονή, αλλά ήθελε κάτι διαφορετικό, δεν ήθελε να περάσει η πρόταση για την αναστολή γιατί είπαμε ότι θέλουμε να μην, ε, μην περάσει αυτού του το, το ύφος αυτού του πολύ. Τέλος πάντων, ε, θα κατέβει η έκθεση στην Ολομέλεια του Απριλίου. Οπότε, σήμερα μπορεί να δοθεί εντολή για έναν τρίμερη διάλογο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια συνεργασία με Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Και ελπίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ο τέλος ακριβώς όπως ήταν και η δουλειά μας στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Στία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ε, καλή δουλειά που έκανε. Τα έχουμε ξαναπεί, οπότε δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους από την ομάδα του ΕΛΚ όχι μόνο εδώ στην ΙΝΤΑ αλλά και στην ΑΦΕΤ που ε, υπέβαλαν την γνωμοδότηση για την ε, ευελιξία που επέδειξαν για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις ε, που να τύχουν ευρεία συνένεση σε αυτή την πρόταση οδηγίας. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη στα πλαίσια της συνολικής ενωσιακής στρατηγικής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα μέτρα που προτείνονται, αυτόνομα εμπορικά μέτρα, θα βοηθήσουν ε, τις χώρες αυτές, ιδιαίτερα για την κατάσταση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, όπως είπε και ο εισηγητής, θέλουμε να ζητήσουμε από την χώρα αυτή να τηρεί τους κανόνες όπως είπε και και εκπρόσωπος δεν μειώνουμε τις προϋποθέσεις αλλά στέλνουμε και ένα σαφές, στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα στήριξης της χώρας να καταλάβει ότι δεν είναι μόνη της, θα τη βοηθήσει η Ένωση στις προσπάθειες αυτές. Αντικειμενική λοιπόν έκθεση, καλή έκθεση, πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθεί ευρέω στην Επιτροπή μας και κατόπιν στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Σκιώδης από ΙΣΙΑ και Άλντε δεν είναι εδώ. Γκουε, επίσης απόν. Ο κύριος Ζανίκ ε, εκπροσωπεί τον κύριο Μπούχνερ. Ευχαριστώ τον εισηγητή που παρουσίασε την άποψη των Πρασίνων. Δεν στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν. Θεωρούμε ότι δεν είναι ισορροπημένη. Η Ευρώπη σε αυτή την περιοχή του κόσμου και στο παρελθόν και τώρα δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τις διάφορες χώρες ο εισηγητή συνέκρινε τη χώρα αυτή με την Ιταλία, αλλά δεν είναι στην ίδια φάση. Η πρόσφατη ιστορία της Ιταλίας δεν συγκρίνεται με την πρόσφατη ιστορία της Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Οπότε υπάρχουν κίνδυνοι αποσταθεροποίησης της οικονομία. πολύ μεγαλύτερη. Δεν στηρίζουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριος Μπορέλη είναι εδώ. Δεν είναι. Οπότε η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα. Δεν θα πω πολλά. Τα περισσότερα ήδη έχουν υποθεί και στις ε, συνεδριάσεις ε, του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε τον Ισηγητή για την υψηλή ποιότητα της έκθεσής του, τη θαυμάσια ποιότητα, όπως και ο Ισηγητής. θεωρούμε οι αυτόνομες προτιμήσεις που δίδονται στα Δυτικά Βαλκάνια είναι κίνητρο για να επιταχυνθεί η τόσο αναγκαία προσπάθεια οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, αλλά το ενδεχόμενο διακοπής είναι επίσης σημαντικό. Υπάρχει ένα θεσμικό πρόβλημα με την τροπολογία για να αντικατασταθούν εφαρμοστικές με κατ εξουσιοδότηση πράξης, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να δρούμε σύμφωνα με τα αυτόνομα μέτρα που έχουμε δώσει ήδη στο Εκουαδόρ και την Ουκρανία. Ελπίζω όμως να υπάρξει ταχύ επίλυση, ούτως ώστε να διατηρηθούν τα αυτόνομα μέτρα και θεωρούμε ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει και το ειδικό θέμα ότι έτσι θα τους δώσουμε και κάποια ενθάρρυνση για να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει και οπωσδήποτε θα ε, ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα τη Κροατία. Ευχαριστώ κύριε Συγητή. Απλώ να πω στον πράσινο συνάδελφο ότι Και αυτά θα πρέπει να τα φροντίσουν πρώτα-πρώτα στο, στο περιβόλι μας. Αυτό είπα, συγκρίνοντας κατάσταση στη Βοσνία με την Ιταλία. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και θα ψηφίσουμε και γι' αυτό στις 10. Να προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ μέχρι τις 10 και στις 10 λοιπόν τα ξαναλέμε για τις ψηφοφορίες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann äh, kommen wir... Frau Πρόεδρος. Συνάδελφοι. Τώρα ήρθαμε στο θέμα υπαριθμών 10 της Μεσικής Διατάξεως. Παρακαλώ, ετοιμάστε τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Τώρα ε, έχουμε το θέμα υπαρτιμών 10, την μακροοικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Okay. Okay. Ε. Yeah. Good. So, wir haben einen Kollegen. Λοιπόν, ένα συνάδελφος δεν έχει την κάρτα του θα την συνυπολογίσουμε την ψήφο του και κάποιος έχει ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό ο κύριος Κάμπελ Ευχαριστώ κάτι διαδικαστικό χθες είχαμε την ακρόαση και θεωρώ ότι τα παρατη... οι παρατηρήσεις ε, της συντονίστριας για την Αμερικανική αρχιτεκτονική ήταν απαράδεκτες γιατί είπε ότι δεν θα ήθελε ποτέ να έχει Αμερικανό αρχιτέκτονα. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα αυτά, τα, αυτές οι δηλώσεις και επιπλέον το EU Trade Insights ήταν συνδιοργανωτής αυτής της ακρόασης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μα δεν είπε αυτό. Ρώτησε αυτό σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να πάρω Αμερικανό αρχιτέκτονα. Έθεσε μία προκλητική ερώτηση σε ένα από τους μας. Εγώ δεν το κατάλαβα καθόλου με αυτή την έννοια. Αυτό θα ήταν ε, ε, λυπηρό. Αλλά μπορούμε να ελέγξουμε την μαγνητοσκόπηση. Πρόεδρος. Την καλέσαμε ως συντονίστρια. και δεν θέλω να επικρίνω τις απόψεις της. Το καθήκον της ήταν να θέτει ερωτήσεις. Και αν δεν μας αρέσουν ε, αυτά που λέει, την επόμενη φορά θα πάρουμε άλλον. Κατά τη γνώμη μου, όλα πήγαν πολύ καλά. Λοιπόν, 10. Μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε 43 τροπολογίες. Θα τις ψηφίσουμε. Λοιπόν, τροπολογία 1 και 2 ταυτόσιμες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 23 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Α, καταπίπτει, 28 Επίσης, και ομοίωση 29 και 30. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Υπαριθμό 34. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 40. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 43. Υπέρ. α, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Ακούσαμε λοιπόν την πρόταση οι επόμενες τραπολογίες να ψηφιστούν ε, unblock, όλες μαζί. Συμφωνείτε, Έλμουτ. Και η 11 και η 19. Α, εκτό από την 11 και 19, διευκρινίζει ο κ. Σόλτ. Εκτό από την 11 και την 19. Συμφωνείτε παρακαλώ όλοι. Πρώτη ομάδα λοιπόν τροπολογιών 4 έως και 10. Ποιος είναι υπέρ. Συνολικά λοιπόν, unblock οι 4 έως 10. Οι κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία υπεριθμών 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Και τώρα παρακαλώ δεύτερη ομάδα η 12 έως 18. Τροπολογία 12 έως 18 μπλοκ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπεριθμού 19. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα η 3 Υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ 7 κατά καμία αποχή και τώρα θα ψηφίσουμε παρακαλώ για το νομοθετικό ψήφισμα. Έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. 29-30 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τριάντα, ναι, τριάντα η ψήφη υπέρ. Και περνάμε λοιπόν στο σημείο 11. Μέτρα κτηροποίησης και σύνδεσης σε ό,τι αφορά την Βοσνία Ζεκουβίνη. 7 τροπολογίες έχουμε. Τέσσερις εξ αυτών, ή μάλλον τέσσερις επιπλέον, τροπολογίες από την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 του εισηγητού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 επίσης του εισηγητή, υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Καταπίπτει 14 και άρα περνάμε τροπολογία υπαριθμών 1 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σε δύο τμήματα. Αφέτ λοιπόν τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη λέει η Κατά. Για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 της Επιτροπής Εκτρικών Υποθέσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Και η τρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καταπίπτει. Και περνάμε λοιπόν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. 32 ψηφί υπέρ. Ναι, ναι, ναι. 32 οι ψήφοι. Υπέρ. Και τώρα να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Έναρξη της ψηφορίας. ψήφι υπέρ, 6 κατά. Ο εισηγητής προτείνει μετά την ψήφιση των τροπολογιών στην Ολομέλεια να αναβλήσει η τελική ψηφοφορία, να ξεκινήσει τη δικασία τριμερού διαλόγου για να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. και προτείνεται να υπάρξει μια διαπραγματευτική επιτροπή. Και αυτή την πρόταση λοιπόν καλούμαστε να ψηφίσουμε. Ποιο συμφωνεί με τη διαδικασία αυτή προκειμένου να δοθεί σχετική εντολή. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε λοιπόν στο σημείο 12 της ημερήσιας διαταξής. Το θέμα της στρατηγικής. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, όσοι φεύγουν από την αίθουσα, παρακαλώ να κάνουν ησυχία. Also, es geht um die Frage der Strategie. Το θέμα λοιπόν της στρατηγικής για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων γενετικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. έκθεση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Μόσκα. Ehm. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Μόσχα. Όπως είπαμε και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αποφασίσαμε στην Επιτροπή μας να λάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, νομοθετική πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρωτοβουλία του Ιουλίου του 2014 εκεί όπου χάστε μια στρατηγική για την ε, προστασία των ε, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές των τελευταίων ετών και κυρίως όσον αφορά τα ψηφιακά οπότε εδώ έχουμε κάποιες προκλήσεις οι οποίες με κάποια μέσα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν είχαμε προσαρμοστεί εις αυτά. Οπότε και γι' αυτό τώρα εκπονήσαμε αυτό το σχέδιο κειμένου. Με αυτό το σχέδιο κειμένου σήμερα θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και να σας επισημάνω ποια είναι τα πλειονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Πόντας επιτροπής. Ξεκινούμε με κάποιες ε, γενικές παρατηρήσεις και το θα πρέπει να δούμε στις λεπτομέρειες ακριβώς πώς διαρθρώνουμε το κείμενό μας. Όσον αυτά τα γενικά, είπαμε ότι βέβαια συμφωνούμε με αυτή την στρατηγική για το ότι τη χάραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε σαν θετικό το ότι δεν θα πρέπει να σβηστεί όλη η προεργασία που έγινε στο παρελθόν. Όλα αυτά να σε σχέση με τη Συμφωνία Άκτα. Και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εκείνα το οποίο είχαν οδηγήσει στη ματέωση της πρωτοβουλία εκείνης. Οπότε έχουμε τώρα μια νέα στρατηγική, σύμφωνα με την οποία τώρα μπορούμε να διοπιστώσουμε κάποια θετικά στοιχεία, δηλαδή να δούμε τι γίνεται με αυτή την στρατηγική. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ως προς τις τρίτες χώρες. πώς θα ε, μπορέσουμε να συμβαδίσουμε τα όσα ισχύουν στο εσωτερικό με τα ισχύουν στις σκήνες της χώρας. Άρα θα πρέπει να λάβουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές πώς αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν. Οπότε και είπαμε ότι κάνουμε τώρα ένα πρώτο βήμα, ούτως ώστε να επισημανθεί το τι είδου ε, συνεννόηση θα πρέπει να γίνει με του εμπορικού ε, ακολούθου, τέλο πάντων με κάποιου ειδικού, για να βελτιωθεί η σχετική ρύθμιση, αλλά και να δούμε και τι κυρώσει θα έχουμε σε περιπτώσει παραβιάσεων. Έχουμε και θετικά σημεία, βέβαια, στην στρατηγική της Κομισιόν. Έχουμε τη διαπίστωση το ότι χρειάζεται μια ηθική δέσμευση όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες. Χρειάζεται περισσότερη συνέπεια όσον αφορά αυτά τα δικαιώματα διανοικής ιδιοκτησίας και τις άλλες πολιτικές, αλλά επίσης θα πρέπει κανείς να δεσμευτεί περισσότερο όσον αφορά τις άλλες χώρες, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, γιατί όλοι φέρουν ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας της προστασίας των δικαιωμάτων. Έχουμε όμως κάποια αρνητικά σημεία. Και δεν προβλέπεται διαφοροποίηση μεταξύ ψηφιακών και υλικών ε, δικαιωμάτων, εμπορευμάτων γιατί θα πρέπει να, για να είναι αποτελεσματική να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Επίσης, άλλο αδύνατο σημείο είναι το τι μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά των χωρών που δεν συμμορφώνονται τόσο πολύ και στο κείμενό μας προσπαθούμε όλα αυτά να τα αποτυπώσουμε. Και έχουμε επίσης προσθέσει και κάποια άλλα στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Εν γέννη, ο στόχος της έκθεσης είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε μια εγγύηση μεταξύ ισορροπίας των κατόχων των δικαιωμάτων και των τελικών χρηστών. Γύρω από αυτόν τον άξονα κινηθήκαμε για την έκθεσή μας και αυτό προσπαθήσαμε και να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας, ένας σύνδεσμος μεταξύ των δικαιωμάτων της μοναδικής ιδιοκτησίας με τις άλλες πολιτικές και να μην ξεχνούμε ότι η παραποίηση σήμερα αφορά κάποια αγαθά τρέχουσες χρήσεις καλλιντικά, φάρμακα κλπ. Οπότε υπάρχουν σημαντικές συνέπειες αρνητικές για την υγεία των πολιτών. Επίσης, εδώ για αυτές τις παραποίησεις απομίσεις έχουμε οργανωμένο έγκλημα το οποίο ασχολείται με αυτό και άρα θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική η οποία και αυτή να συνδεθεί με τις πολιτικές μας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Και βέβαια μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά τα οποία διακυβεύονται εδώ και όπως λέγαμε χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ ψηφιακών και μη ψηφιακών επίσης ότι θα πρέπει το συνεμότερο δυνατόν να γίνει μια προβληματική για να συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος τα θέματα, τα προβλήματα αυτά. Επίσης επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να συναρθούν κάποιες συνθήκες διαφορετικών ε, ειδών γιατί Έχουμε πρώτα πρώτα την καταπολέμηση της παραποίησης, την ε, προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, χρειάζεται να εμπλακούν εδώ περισσότερο, περισσότεροι, ας πούμε να συνεργαστεί η ΙΚΑΝ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκτός από τις επιχειρήσεις, γενικότερα να συμμετάσχουν και οι τρίτοι. Φερρυπίν, εννοούμε τις τράπεζες. Γιατί υπάρχουν έτσι μηχανισμοί που μπορούν να εξασφαλίσουν τήρηση του νόμου αλλά και κυρώσεις. Οπότε θα πρέπει τώρα να δούμε πώς να τον έχουμε πιο υψηλά πρότυπα τα οποία θα τάξουμε Οπότε αυτό θα πρέπει να ισχύει όπου και όποτε κάνουμε διαπραγματεύσει με τι τρίτε χώρε. Και γι' αυτό σα λέω ότι χρειάζεται να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Στο ότι κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται κάποιε εμπορικέ συμφωνίε θα πρέπει το κεφάλι που αφορά την πνευματική ιδιοκτησία να το θεωρούμε πάρα πολύ βασικό. Επί του οποίου δεν θα, δεν θα είναι απλώ μια προσθήκη, ένα παράρτημα που θα αποσαρτάται, αλλά θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα του σώματος της συμφωνίας και άρα εκεί θα έχουμε την προστασία των δικαιωμάτων αλλά και των γεωγραφικών ενδείξεων. Επίσης, τελευταίο, θεωρούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Παρατηρητής όσον αφορά τις παραβιάσεις της και την κυβερνητική εκκλησία θα πρέπει αυτός να έχει την απαραίτητη πρικοδότηση και πόρους ούτως ώστε να μπορεί να παράσχει αυτές τις εγγυήσεις ότι θα επιτελέσει το έργο του και επίση θα πρέπει να έχει ανεξαρτήσει όσον αφορά τη διαχείριση του έργου του και εδώ θα βάλω μια τελεία αλλά βέβαια είμαι πρόθυμο να συζητήσω ότι μπορούμε να πούμε για να βελτιώσουμε την έκθεση. Πρόεδρος. Τώρα η Σκιώδης. Ο κύριος Βίζας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την θαυμάσια εργασία πρώτα απ' όλα. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση των σκιωδών που νομίζω πως ήταν πολύ παραγωγική. Εκφράστηκα επί της εκθέσεως και επί δύο-τριών σημείων επί των οποίων έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Επαναλαμβάνω, θεωρώ πολύ καλή την έκθεση. Και από ορισμένε απόψεις είναι πιο πλήρη και από την ίδια την πρόταση της Επιτροπής. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και η ομάδα μου δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να στηρίξει αυτή την έκθεση. Παρ' όλα αυτά, να ασχοληθώ με τα σημεία. Τα συζητήσαμε χθε, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικά να τα ε, θέσω υπόψη και τη Επιτροπή. Για να τα συζητήσουμε. Στο σημείο 12 της έκθεσης η συγγήτρια λέει οι, τα, οι συμφωνίες TRIPS να είναι πιο ευέλικτες. Έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι αποδυνάμωση των διατάξεων το οποίο δεν θα ήταν ε, Ε, δεν θα ήταν κάτι που θα ενίσχυε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Όμως ε, η συγγήτρια μας είπε ότι δεν είναι η πρόθεσή της, αλλά θα υποβάλουμε τροπολογία να το διευκρινίσουμε. Για το σημείο 20 λέει ότι η Κομισιόν θέλει να έχουν ε, τη δυνατότητα οι τράπεζες να τιμωρούν απευθείας ε, τις απάτες ε, στο ίντερνετ. Ε, δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να εφαρμόζουν κυρώσεις. Ούτε μπορούν ούτε είναι αυτές που θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις. Αυτό είναι το πιο μέχο για μας. Άλλο σημείο για το οποίο έχω αφιβολήσει είναι το 22. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης υπογράψει τις συμφωνίες που αναφέρονται. Οπότε Εάν δεν τις έχουν προσυπογράψει τα κράτη-μέλη, δεν μπορούμε να ζητάμε από τρίτες χώρες να επικυρώσουν. Δεν μπορούμε επίσης να ζητήσουμε άλλοι να εφαρμόσουν το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν. Και να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με τις χώρες της Ένωσης. Άρα χρειάζεται μια κάποια αναλογικότητα όσον αφορά τις απαιτήσει που θέλουμε να επιβάλλουμε σε αυτές τις χώρες για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες που να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα να επικυρώσουν τις συμφωνίες αυτές και να ενθαρρύνουμε τις χώρες που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα να εργάζονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές αυτών των συμφωνιών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως υποτιμώ τη θαυμάσια εργασία της κυρίας ε, Μόσκα και παραλαμβάνω ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα για να την εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Η ΕΜΑ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ την εισηγήτρια, το μεγαλύτερο τμήμα τη έκθεση το στηρίζουμε και όπω είπε και η συγγήτρια στην αιτιολογική τη έκθεση και όπω είπα και εγώ στην ε, συζήτηση χθε, είναι περιορισμένε οι ενέργειε που έχουν γίνει για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό και παρά τι αλλαγέ ε, στην τεχνολογία και την κοινωνία που είχαν τεράστιε επιπτώσει σε τέτοια θέματα. Άρα, να ασχοληθώ με αυτό που λέει και η έκθεση και η ανακοίνωση τη Επιτροπής αυτό που συζητάμε να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ των ε, συμφερόντων των δικαιούχων και των χρηστών. Σε διάφορα σημεία της έκθεσης το λέμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εφόσον ε, διαμορφώνουμε πολιτική για να επιτύχουμε αυτή τη συμφωνή, την ισορροπία. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε μετά αυτά που συνέβησαν με την άκτα για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ήδη εξέφρασα τις ανησυχίες μου όταν συζητήσαμε την άκτα και θα ήθελα να μου πει η συγγήτρια τι μπορούμε να επιτύχουμε από την αποτίμηση τη διαδικασία άκτα. Πρέπει πραγματικά αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Πρέπει να αυξηθεί η ευαισθησία του κοινού για το ότι δεν εφαρμόζονται τα δικαιώματα διανοτικής ιδιοκτησίας. Κάτι άλλο που επίσης λέει η ιδεολογική σκέψη AIDS. Πρέπει να έχουμε υπόψη όχι μόνο τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τις ε, επιχειρήσεις μας και τους δημιουργούς μας, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και την ίδια την δημιουργικότητα. Εάν δεν αμείβονται οι δημιουργοί για την εργασία τους, θα σταματήσει η δημιουργία. Και, και οι χρήστες λοιπόν δεν θα έχουν ε, την ποικιλία διανοητικών προϊόντων που είναι η περηφάνεια της Ευρώπης. Συμφωνώ με την εισηγήτρια να μας πει περισσότερα η Κομισιόν για πόσοι πόροι θα χρειαστούν για να επιτύχουμε τους στόχους που θέλουμε για την ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων. Και ελπίζω να μας πει η Κομισιόν σήμερα τι θα χρειαστεί, πόσο προσωπικό, ποιες περαιτέρω προτάσεις για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη και για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη για συντονισμένη προσπάθεια. Και αυτό σχετίζεται και με τα τελωνία και την επιτήρηση της αγοράς. Να είμαστε λοιπόν ε, συντονισμένοι και όχι να κάνουμε όλη την ίδια δουλειά. Ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Αποτελεσματικός διάλογος με τις χώρες προτεραιότητας και περιφέρειες προτεραιότητας. Και αυτό πολύ σημαντικό. Θα παίξει ρόλο κλειδί στο πώς θα προσεγγίσει η Κομισιόν το θέμα αυτό. Πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις με τις χώρες αυτές να έχουν υψηλές προδιαγραφές για την προστασία εντός των χωρών αυτών των ε, δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να εργαστούμε από αυτού. Θα στηρίξω λοιπόν αυτή την έκκληση να συνεχίσει η Επιτροπή να αυξάνει τις προσπάθειες, να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτω ώστε να βελτιώσουν τα συστήματά τους προστασίας. Τεχνική βοήθεια μπορούμε να τους δώσουμε και κατάρτιση. Και επίσης μπορούμε να εξαγάγουμε τέτοια μέτρα προστασίας. Για να το κάνουμε αυτό, τα κράτη-μέλη πρέπει τα ίδια να επικυρώσουν τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτή τη σύμβαση, για παράδειγμα, για τα σήματα κατά τεθέν. Πώς θα μας πάρουν σοβαρά όταν τους καλούμε και καλούμε και τον ΜΠΟΕ να προτείνει τέτοιες συμφωνίες, εάν εμείς δεν έχουμε επικυρώσει παρόμοιες. Συμφωνώ λοιπόν τις εκκλήσεις. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη. Να γίνει αυτό επιτέλους. Ανησυχώ λιγάκι όσον αφορά την παράγραφο 22, το είπε και ο συνάδελφος Φίσας, που λέει να προσταθούν και άλλες συμβάσεις στις υπάρχουσες 27 για να μπορούν οι χώρες να συμπεριληφθούν στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, ΣΥΝ. Αυτή η συμφωνία θέλει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η καλή διακυβέρνηση στον τομέα αυτό. Αν ακολουθήσει η πρόταση, αν ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόταση θα γίνει ε, υπερβολικά περίπλοκο όργανο. Αντί λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό, να βάλουμε ίσως μια αναφορά σε άλλους τομείς της έκθεσης με πιο κατηγορηματική διατύπωση, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα μπορούσαμε λοιπόν ίσως να συμφωνήσουμε σε μια διατύπωση. Και τέλος, τέλος, να ασχοληθώ με την παράγραφο 36. Καλεί την Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες για την ε, επέκταση της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα. Δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό. Θα το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο μετά το πράσινο, την πράσινη βίβλο της Επιτροπής. Το πράσινο έγγραφο. Να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και ε, καλό την Κομισιόν να περιμένει πριν πάρει περαιτέρω μέτρα αλλά βεβαίως προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών. Γενικά συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η προστασία και ελπίζω να καταλήξουμε σε κοινή θέση και να είναι πολύ στεναρή αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έλλη μου το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ Θέλω να αντικαταστήσω την Άννα Μαρή που είναι σκιώδης από την ομάδα μας και δυστυχώς σήμερα έπρεπε να παρευρεθεί στην Ολλανδία που έγινε εκλογέ στην περιφερειά της. Γι' αυτό λοιπόν και παίρνω το λόγο εξ ονοματός της. Θέλω να ευχαριστήσει λοιπόν τον εισηγήτρια για την προσέγγιση της, για την έκθεση την οποία κατήρτισε. Να τονίσει επίσης ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στην έκθεση της ε, κυρίας ε, Μόσκα, με τις οποίες συμφωνούμε, αλλά θέλουμε να προσθέσουμε και κάποια στοιχεία. Μας επενθυμίζει λοιπόν η συνάδελφος ότι θα πρέπει να διδαχτούμε από τα παθήματα της Συμφωνίας Άκτα και το θα πρέπει να λάβουμε τα στοιχεία αυτά υπόψη μας. Επίσης, η κυρία Μόσκα επιμένει για μια πιο εκδεδομένη συζήτηση για τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα θα διτεθούν στο κοινό. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να αφήσουμε την υγεία στα χέρια της αγοράς. Η αγορά είναι για να βγάζει κέρδος, αλλά όχι για να την εμπιστευόμαστε. Δεν μας αρέσει λοιπόν ε, το σημείο 27 που αναφέρεται τα φάρμακα που πολλούνται και μεταπολούνται σε τρίτε χώρε. Θα πρέπει να είναι πάντα σαφέ οι προτεραιότητε. και δεν είναι σαφέ. ότι τα νέα αντιβιωτικά που χρειάζονται για παράδειγμα δεν αναπτύσσονται και οι φαρμακευτικές εταιρείε διαλέγουν ποια φάρμακα θέλουν να εξελίξουν. Και επίσης ε, στο σημείο 31 αναφέρονται τα θέματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησία. Ε, αναφέρονται διάφορες στοιχείες υποθέσει από το πατήριο στο Μόναχο. Στο 39. Εδώ είμαστε πιο επιφυλακτικοί από ότι οι άλλοι για τη Σύμφωνη ελευθερίου εμπορίου. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να είναι τόσο σημαντικό στοιχείο. Και δεν βλέπουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παίζει ρόλο όπω αναφέρεται στο σημείο 43, σε θέματα επίλυση διαφορών. Αυτό θα πρέπει να είναι εθνική αρμοδιότητα. Τέλο, η Αν Μαριμέρ τονίζει ότι θα πρέπει να ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να τον τονίσουμε ότι οι νέες εφευρέσεις θα πρέπει να ωφελούν και την κοινωνία και τους πολίτες. Ε, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα θα πρέπει να το δίνουμε προτεραιότητα στην κοινωνία και όχι στην αγορά. Γιατί η κοινωνία συμβάλλει στους όρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε ό,τι αφορά τις σχολές, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, αλλά παρέχει και τις σχετικές υποδομές που χρειάζονται. Είναι λοιπόν λογικό το όφελος να το έχει η κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πιο πολύ και όχι να ακολουθήσουμε μια ενοποιημένη ομοσπονδιακή προσέγγιση. Ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή γιατί ασχολήθηκε με ένα περίπλοκο θέμα. Εδώ και πολύ καιρό δούμε, να δούμε, να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ προστασία τη ε, καινοτομία, τη ε, δημιουργία αλλά και τη ε, δυναμική εξέλιξη τη κοινωνία και να αποφύγουμε η προστασία να καταστεί ένα μονοπόλιο. Και αυτό το οποίο προσφέρει ενδιαφέρον είναι αυτή η διάκριση μεταξύ των υλικών αγαθών και δικαιωμάτων και των ψηφιακών γιατί μιλούμε για συνεχή εξέλιξη σήμερα και ακόμα και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι σε αυτά τα δικαιώματα δεν έχουν καταλάβει 100% τι ισχύει και τελικά τι πρέπει να συνεπάγεται η προστασία. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρό το τι, ποια, ποια είναι η ευθύνη των ε, παρόχων υπηρεσιών ε, ίντερνετ. Ακριβώς αυτό ήταν το αντικείμενο της ε, άκτα που δεν ευδοκίμησε. Ακριβώς και εμείς αυτό θέλουμε να το πούμε στην εισηγήτρια και έχουμε το άρθρο 19 εκεί όπου μας ε, τονίζει ότι υπάρχει ευθύνη από πλευράς των ε, ε, παρόχων αυτών και όμως θα πρέπει να το κοιτάξουμε και να το ρυθμίσουμε ενδελεχέστερα. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ουδετερότητα του δικτύου. Ευχαριστώ, λέει ο Από το e δεν έχω σκιώδη. Δεν έχω λοιπόν κανένα άλλο που να ζητάει το λόγο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Πιέτρο Βελάσκο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε σε πρώτη φάση να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για τον ανοιχτό πνεύμα που έδειξε και την, τον διαφανή τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και προετοίμασε την έκθεση αυτή. Μας άκουσε με μεγάλη προθυμία και στη συνέχεια έκανε πολύ καλή δουλειά και έτσι καταλήξαμε σε αυτή την πολύ λεπτομερή αξιολόγηση. Σημειώνουμε λοιπόν τα πολλαπλά στοιχεία της έκθεσης αυτής που εξετάζει με θετικό τρόπο τη στρατηγική. Μετά από την θετική αξιολόγηση και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Υπάρχει ισόρροπη προσέγγιση σε ό,τι αφορά και τα διάφορα διφατικά σε κάποιες περιπτώσεις συμφέροντα. Αυτό ανησυχεί καθημερινά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φαντάζομαι και το Κοινοβούλιο η σημασία της εναρμόνισης της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής δικτυσίας και των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποστήριξη για το έργο μας σε ό,τι αφορά την εντοπισμό των χωρών προτεραιότητας, τη συμφωνία για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το παρατηρητήριο. που θα πρέπει να έχει τους σπόρους ε, και τις δυνατότητες να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει. Συνεχιζόμενη προώθηση της επιβόλησης των δικαιωμάτων γενετικής ιδιοκτησίας, αυτό ασφαλώς κοστίζει χρήματα χρήματα που δεν έχει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου στη διάθεσή τη. άρα πρέπει να συντονιστούμε με του συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση ανάπτυξη και ασφαλώ να έχουμε την υποστηρίξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αναγνωρίζεται επίση η περιπλοκότητα του θέματο των ε, φαρμάκων που ξεπερνάει κατά πολύ το θέμα των δικαίωματων διανοητική ιδιοκτησία. Μεγάλη τμήμα τη συζήτηση εστιάζεται φυσικά σε αυτά, άρα το θέμα είναι πολύ πιο πολύ σύνθετο. Τη σημασία που δίνεται σε μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για να προωθηθούν τα πρότυπά μα σε τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να ζητάμε από άλλου να κάνουν αυτά που δεν κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Κάτι που δεν αναφέρθηκε σήμερα, αλλά η σημασία να συνεχίσουμε να προωθούμε τα θέματα αυτά σε πολυμερή φορά όπως ο ΠΟΕ η σημασία της διανοτικής ιδιοκτησία σε συμφωνίες ελευθερού εμπορίου. Αυτό στη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής στις νέες συμφωνίες με την ε, Νότια Κορέα, με τον Καναδά. Έχει αποτελέσει κεντρικό ζήτημα και έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, την υποστήριξη του διαλόγου για θέματα δυνατικής ιδιοκτησίας αυτό ίσως να το θεωρείτε κάποιες φορές ε, ήπια, διπλωματία. Μία άσκηση που γίνεται με, ευρωπαϊκούς, με ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε τέτοιες χώρες μέσω διαλόγου, μέσω επικοδομητικής συζήτησης με τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών που αποτελούν χώρες προτεραιότητες και για τη συνεργασία με τις περιφερειακές ομάδες. Σημειώσαμε με ενδιαφέρον κάποιες προτάσεις που ξεπερνούν κατά κάποιο τρόπο αυτά που περιλαμβάνονται στη στρατηγική. Για παράδειγμα, η σύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και παραβίασης δικαιωμάτων γενετικής ιδιοκτησίας εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν έχει περιορισμένο ρόλο, δεν υπάρχει κεκτημένο. Η ανάγκη για πιο ενεργό ρόλο στο ICANN στο σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών σε ό,τι αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, ΣΥΝ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχουμε κοιτάξει κατά την προετοιμασία της στρατηγικής. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, αλλά αν προτείνει κάτι τέτοιο το Κοινοβούλιο, να εξετάσουμε αυτό το θέμα πιο εντελεχώς, εμείς θα το πράξουμε. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Και επίσης ε, μεγαλύτερη χρήση του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Δεν είναι απλά τα πράγματα γιατί στο σύστημα του ΠΟΕ αυτό το σύστημα επίλυσης διαφορών σημαίνει τη μεταφορά σε νομοθεσία των διατάξεων αυτών στις τρίτες χώρες. Αυτό γίνεται θεωρητικά, αλλά τα προβλήματα συνήθως προκύπτουν κατά την εφαρμογή των νόμων. Για το θέμα τώρα των πόρων. Καταγράφουμε τις δράσεις εφαρμογής και αυτό το κάνουμε εντατικά. Την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, θα παραστώ σε ένα διάλογο για τα τεχνητικά δικαιώματα στην Τουρκία και σύντομα θα δημοσιεύσουμε τον κατάλογο των χωρών προτεραιότητας στο τρέχον έτος. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, συνεργαζόμαστε με τους εμπλεκόμενους φορείς και διοργανώνουμε ήδη μετά τη δημοσίευση της στρατηγικής ε, μία συνάντηση με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς για να συζητήσουμε θέματα πρόσβασης σε φάρμακα. Έχουμε πολύ καλές επαφές με κάποιες ΜΚΟ. Και τέλος υπάρχουν κάποιες προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στη σύσταση που δεν σχετίζονται άμεσα με τις εμπορικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, όλο αυτό το θέμα με τους ε, ενδιάμεσους σε ό,τι αφορά το μνημόνιο συνεννόησης με σημεία πώληση στο διαδίκτυο φαρμάκων παραποιημένων. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονταν στο σχέδιο δράση του Επίτροπου Μπαρνιέ από τη Γενική Διεύθυνση Αγορά, το οποίο πλέον έχει περάσει στα αρμοδιότητα τη ε, γενική διεύθυνση Grow ε, και θα του και εξετάζουν τι προτάσει αυτέ. Αλλά μέτρα συνεπάγονται νομοθεσία, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων στι ε, τράπεζες. Αυτό δεν ήταν ο σκοπό μα ο σκοπός μιας στρατηγικής τέτοιας έχει μεταβιβαστεί αυτό ασφαλώς και έχει μεταφερθεί στους αρμόδιους ε, συναδέλφους σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα μονοπόλια στον τομέα των φαρμάκων. Αυτό σχετίζεται πιο πολύ με θέματα ανταγωνισμού και όχι τόσο πολύ με τη δική μας στρατηγική για τα δικαιώματα διανέζικη συντεκτησία. Σημειώνουμε επίσης την επιθυμία του Κοινοβουλίου να εισακουστούν οι αξιώσεις μας και οι ανάγκες μας, γιατί όλα αυτά συνεπάγονται μεγάλη ανάγκη σε πόρους, είναι πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρε ως διαδικασίες. Δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό στο, στις κορυφαίες 10 προτεραιότητές μας. Αλλά για επιτραμμένη σε θέματα διανοητικών δικαιωμάτων στην κεντρική και στην ανατολική Ασία και στη Λατινική Αμερική ή και στην Ασία. Προσπαθούμε να βρούμε και άλλες λύσεις, να δημιουργήσουμε μια σχετική ε, υπηρεσία στην Κίνα. Ψάχνουμε λοιπόν και να ζητούμε λύσεις και στα πλαίσια του παρατηρητηρίου, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα πόρων. Είμαστε λοιπόν ε, πρόθυμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και να συνεχίσουμε να σημειώνουμε το οτιδήποτε προτείνει το Κοινοβούλιο για τη στρατηγική μας, γιατί είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία αυτή. Η στρατηγική θα συνεχίσει να εξελίσσεται τα επόμενα πέντε χρόνια και πάντα. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε καινούργιες ιδέες, νέες ιδέες, καινούργια μέτρα. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η συγκεκριά, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για όλες τις ε, παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να σας καλύψω σε σχέση με αυτό που μου είπατε. Κοιτάξτε, πρώτα πρώτα. Ήδη έχω φτιάξει κάποιες ε, τροπολογίες επί τη βάση των όσων αυτή τη βδομάδα μου έχετε πει. Και νομίζω ότι ήδη βελτιώνουν τις διατάξεις τις οποίες τώρα σχολιάσατε. Ό,τι ό,τι δεχόταν δηλαδή διασάφηση. Για να δούμε τώρα συγκεκριμένα. Πρώτα πρώτα έχουμε το 12. Ε, όπως είπε κάποιος συνάδελφος από το ΕΛΚ που αφορά την πιο ευέλικτη ε, εφαρμογή της συμφωνίας TRIPS. Ναι, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις τροπολογίες, γιατί δεν ήταν σαφές το τι πρέπει να γίνει και άρα θα πρέπει να βρεθεί ο πιο σωστός τρόπος για να έχουμε την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της TRIPS ανάλογα με την χώρα που αφορά. Ναι, φυσικά θα έχετε βελτίωση η διατύπωση εδώ τώρα. Κάτι άλλο το οποίο είπαν περισσότεροι συνάδελφοι και αναφέρθηκαν στην τραπεζική παρέμβαση. Όπως είπα και εγώ στην αρχική μου εισηγήση ότι θα πρέπει να δούμε ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να εμπλακούν εδώ, ούτως ώστε να υπάρξει κατανομή της ε, ευθύνη σε περίπτωση παραβιάσεων. Να δούμε πώς θα θωρακίσουμε το μηχανισμό κάθε φορά που κάποιοι προσπαθούν να εμπορευτούν, να πωλήσουν τέλο πάντων παραποιημένα εμπορεύματα. Να έχουμε κάποιες πρωτότυπες εφάνταστες λύσεις και αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα ούτω ώστε να μπορέσουμε να ανασχέσουμε αυτέ τι παραβιάσει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα για το σύστημα προτιμήσεων, συν εγώ δεν θέλω να χειροτερεύσω την κατάσταση, να κάνω λιγότερο ευέλικτη την κατάσταση στις χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία να μην έχουμε πιο επαχθεί διαδικασίες χωρίς εκείνες από όσους έχουμε εμείς εδώ. Πάντως βέβαια είναι σωστά αυτά που μας ανέλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι θα πρέπει γίνει. Γιατί μια που μιλούμε τώρα για παραβίαση δικαιωμάτων μοναδικής ιδιοκτησίας με την παραποίηση, έχουμε περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Άρα είναι καθήκον μας όπως λέμε για προστασία του περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απασχόλησης, θα πρέπει να δούμε σε ποιες περιπτώσεις η παραποίηση και η απομίμηση έχει τέτοιες συνέπειες για την ζωή των πολιτών και σε τρίτες χώρες. Άρα θα πρέπει να διερευνήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε προς αυτό το μέτωπο για τις τρίτες χώρες. Τώρα, όσον αφορά τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, έχουμε το θέμα του copyright. Οπότε και στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μας έχει, κρατά καλά συζήτηση όσον αφορά κάποιου είδου ε, εσωτερικές ρυθμίσεις. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να προδικάζει το αποτέλεσμα αυτής της προβληματικής. Απλώς η μία ρύθμιση να μην αντιβαίνει στην άλλη. Να μην υπάρχει αντίφαση. Θα πρέπει εκ παραλίλου να προχωρούν αυτές οι δύο συζητήσει και ρυθμίσει τρώσαν όλα τα φάρμακα. Συμφωνώ 100% για το ότι τα φάρμακα θα πρέπει να διέπονται από κάποια ρύθμιση, μια που δεν είναι απλώς θέμα αγοράς, είναι θέμα υγείας του κόσμου. Αλλά τόνισα στην έκθεση ότι θα πρέπει να επισημαθούν οι τομείς όπου θα μπορούσε να υπάρχει διαφοροποίηση της τιμολογικής πολιτικής. Και έτσι να αποφύγουμε στη συνέχεια να έχουμε κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι θα επιφέρουν στρέβλωση ή να δώσουμε το δικαίωμα σε κάποιους να εκμεταλλευτούν και να εισχροκερδίσουν. Μιλούμε για κάποιες χώρες όπου υπάρχουν διαφορετικές τιμές. Εκεί κυρίως θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Εκεί θα αναφύουν αυτές οι δυσκολίες σε σχέση με τα φάρμακα. Και σας ξαναλέω, το θέμα δεν είναι οικονομικό. Και δεν προτείνω γι' αυτό την διαφοροποίηση. απλώ σας είπα ότι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην καταλήξουμε σε καταχρηστικές ε, συμπεριφορές. Α, για το παρατηρητήριο τώρα. Όχι, δεν λέμε να φτιάξουμε καινούργιο παρατηρητήριο. Ας αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο ήδη τώρα λειτουργεί. Αλλά να το προκοδοτήσουμε καλύτερα. Ακριβώς γι' αυτό σας λέω. Χρειάζεται συντονισμός από την Επιτροπή. Δεν είναι θέμα κρατών μελών χρειάζεται συντονισμός και αυτός να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό αφορά και τις ρυθμίσεις για τα τελωνία. όσον αφορά τη σχέση μας με τις τρίτες χώρες. Δεν το είπα στην αρχή, αλλά το αναγράφω στην έκθεση. Το ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε τις διμερείς επαφές παράλληλα με τις ε, πολυμερείς και συνέχεια να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και στι διμερείς συμφωνίες επανέρχομαι όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Πάντως η προτεραιότητα δίνεται στα φόρατα πολυμερή και στι συμφωνίε τη πολυμερή. Επίση, ο πρώτο του του Ιντερνετ, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είδατε ότι δεν έπιασε τόπο το άκτα στην προηγούμενη θητεία και τελικά θα πρέπει και το είπα περισσότερες από μια φορές να έχουμε όσο γίνεται πιο ισορροπημένη προσέγγιση δεν θέλω να επιβαρύνουμε περισσότερε ευθύνε σε αυτούς τους παράγου υπηρεσιών Ιντερνετ. Να υπάρχει κάποιο είδου υπόμνημα μνημόνιο κατανόηση. Ό,τι ρυθμίσει υπάρχουν τώρα επιδέχονται βελτίωση. Γιατί μπορούν να εμπλακούν περισσότεροι για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό που επιδιώκουμε. Να επισημανθούν οι περιπτώσει των παρανομιών, των παραβιάσεων. Και να ρίχνουμε, να μπλοκάρουμε αυτονούν που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις τους ιστότοπους. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην ήδη κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Νομίζω ότι θα, πρέπει να τα λάβει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι να εκπονίζει μια στρατηγική όσο γίνεται πιο αποτελεσματική. Και σε σχέση με το άκτα θα πρέπει να δούμε πώς θα εμπλακούν περισσότερο οι πολίτες να έχουμε ας πούμε μια πρωτοβουλία η οποία και να είναι αποτελεσματική αλλά και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι για το συμφέρον τους και όχι εναντίον του. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, κλείνουμε αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης. Προθεσμία για τροπολογίες 23 Μαρτίου 5 ώρα το απόγευμα. 23 Μαρτίου 17 η ώρα. Στην επόμενη συνεδρίασή μας, 13-14 Απριλίου, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και στις 7 Μαΐου θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο σημείο 13 της σημερινής διάταξης. Είναι η γνωμοδότησή μας για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια, και την στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια προθεσμία τροπολογιών ήταν 26 η Δευτέρου. Έχουμε 83 τροπολογίες. Οπότε να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Κιώδης και όλους τους άλλους συναδέλφους για μια πολύ επικοδημητική συνεργασία που είχαμε. Συνεργασία έντονη για αυτή τη γνωμοδότηση για την ε, Ήτρε που είναι επί της ουσίας αρμόδια με εισηγητή τον κύριο Σαουγκάρδας και την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε είχαμε καταλήξει ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευρύ ότι θα επηρεάσει πολλά θέματα της ενεργειακής ε, καθημερινότητας και των χωρών μας και των τρίτων χωρών, γιατί υπάρχουν και οι διεθνείς πλευρές της ενεργειακής ασφάλειας που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Ότι λοιπόν η ανακοίνωση επί της οποίας γνωμοδοτούμε στα πλαίσια της έκθεσης δημοσιεύθηκε πριν από ένα χρόνο Εφόσον θα ψηφίσουμε στις 7 Μαΐου, αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί ένα χρόνο μετά την ε, θέση της Επιτροπής και μεταξύ. έχουν υπάρξει πολλές άλλες ε, τοποθετήσεις και αυτές οι ιδέες για μια ενεργειακή ένωση με πέντε κέντρα βάρου ε, που υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σεύκοβιτς. Και έχουν ανακοινωθεί και άλλες δύο πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα η συμβολή της Ένωσης στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα το Δεκέμβριο που σχετίζεται με την Ενεργειακή Ένωση και την Ενεργειακή Συνεργασία και το δεύτερο ο στόχος 10% διασύνδεση που θα εξετάσουν τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετάδοσης. Είναι λοιπόν ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί σφαιρικά το Κοινοβούλιο. Δεν είναι τόσο εύκολη κατάσταση λοιπόν. Και γι' αυτό ενέκρινα την πρόταση του ΕΛΚ ε, αμέσως να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Να αναβάλουμε για τον Απρίλιο. Για να έχουμε λίγο χρόνο για να εξετάσουμε και αυτά τα θέματα που ενέκυψαν εντωμεταξύ. Να σκεφτούμε δηλαδή μήπως θα πρέπει να συμπληρώσουμε με προφορικές τροπολογίες αυτές τις 83 τροπολογίες για να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα ακριβώ που έχουν προκύψει. Η γνωμοδότησή μας αφορά όλα τα θέματα της Επιτροπής μας, οικονομική συνεργασία δηλαδή για την παραγωγή ενέργειας, ε, τις πρώτες ύλες, ε, την ε, καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πολλές λοιπόν τροπολογίες για πολλά θέματα. Και έχει υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ εμού και των σκιωδών για το όλες αυτές οι τροπολογίες που αφορούν διάφορα σημεία της αρχικής γνωμοδότησης, πώς μπορούμε να τις αναδιατάξουμε ούτως ώστε να τα συμπεριλάβουμε όλα και παρόλα αυτά να έχει συνοχή η πρότασή μας. Ήδη λοιπόν έχουμε μια σειρά από συμβαστικές τροπολογίες που θα τις συζητήσουμε περαιτέρω με τους κοιόδης που αφορούν πώς θα ληφθεί υπόψη η ενεργειακή ασφάλεια και η παραγωγή ενέργειας στις εμπορικές συμφωνίες. Θέλουμε να τονίσουμε περαιτέρω το σημείο αυτό, περισσότερο. Οι τροπολογίες μιλούν επίσης για την διαφοροποίηση των τρόπων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ένωση και στη συνεργασία μας με τρίτες χώρες για να μειωθεί η εξάρτηση. Πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις ακριβώς για τη διαφοροποίηση, και την τροποποίηση του ενεργειακού μείγματος για να συμμετάσχουν περισσότερο οι εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Αυτό περιμένουμε και από τη δεύτερη ανακοίνωση της Κομισιόν. Πώς λοιπόν η ενεργειακή ασφάλεια θα βοηθήσει την ε, καταπολέμηση της αλλαγής κλίμακος, κλίματος, αλλά και ε, κοινωνικές πλευρές του θέματος. σχετίζονται όλα αυτά με την εξωτερική πολιτική και την εξωτερική οικονομική πολιτική της Ένωσης. Τέλος, θεωρώ ότι η ενέργεια είναι πολύ περίπλοκο θέμα και γι' αυτό δεν πρέπει τόσο μονομερός να ασχολούμεθα με την ευρωπαϊκή κατάσταση όπως κάνει η έκθεση στην Ήτρε αλλά να σκεφτούμε και πώς θα συμβάλλει η Ένωση στην παγκόσμια σταθεροποίηση της ενέργειας, ούτε ώστε να έχουν οι πολίτες παντού ενέργεια και τονίζω ότι πιστεύω ότι η πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και η Επιτροπή μας πρέπει να το αναφέρει. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τη στήριξή της και προσβλέπω στην περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και ήδη την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε άλλη μια συνάντηση με τους σκιώδεις για να συνεχίσουμε την προσπάθεια ε, εξέβρεση συμβασμών γιατί μετά θα έχουμε τη διακοπή του Πάσχα οπότε πρέπει να εργαστούμε σύντομα. Ευχαριστώ Ισκιώδης τώρα λέει ο Πρόεδρος για το ΕΛΚ ο κύριος Σιένφελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, γιατί ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για αυτόν να ολοκληρώσει το έργο του, δεδομένου του ότι κατατέθησαν και 83 τροπολογίες. για να φτιάξει συμβιβασμούς με περιεχόμενο αποδεκτό δεδομένης και της δυσκολίας ε, που προέκυψε από το γεγονός ότι το αρχικό κείμενο της γνωμοδότησης δεν θα μπορούσε να γίνει αποτεκτό. Αλλά και πολλές από τις τροπολογίες ε, που κατατέθησαν δεν θα περνούσαν. Θεωρώ ότι πολλές από τις ε, τροπολογίες δεν αναφέρονται καν στο έγγραφο. Από ό,τι φαίνεται κάποιοι έθεσαν ε, ζητήματα όπως η πολιτική για το κλίμα, για την ενέργεια, γενικά όμως. Και το συγχαίουν αυτό με την στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. Όχι μία παγκόσμια στρατηγική, ούτε για την, για την Ευρώπη συγκεκριμένα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική για το κλίμα θα πρέπει να είναι οριζόντιο έγγραφο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έτσι γίνεται συνήθως, αλλά οι πολιτικές για στρατηγικές θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες ε, πολύ συγκεκριμένα έγγραφα συνεκτικά και στοχευμένα που θα αναφέρονται μόνο στους συγκεκριμένους στόχους, μόνο στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. που χρειάζονται για την στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αν στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής για την ε, ενέργεια και το κλίμα προσπαθούμε να βάλουμε γενικές ιδεολογίες και κάποια γενικά σχόλια, δεν θεωρώ ότι θα καταλήξουμε πουθενά. Και οι πιο πολλές από τις τροπολογίες προτείνουν να εισαχθούν στο έγγραφο αυτό στοιχεία τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά να κάνουν τίποτα με την ενεργειακή ασφάλεια για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γεγονός ότι κατάφερε ο εισηγητής να φτιάξει αυτούς τους επτά συμβιβασμούς, να τους πετύχει αυτούς τους επτά συμβιβασμούς ήταν αξιοθαύμαστο. Τώρα λοιπόν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με τους συμβιβασμούς αυτούς να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Και τώρα επιτρέψτε μου να είμαι πιο συγκεκριμένο να αναφερθώ σε συγκεκριμένα στοιχεία, σε συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί που μπορεί να γίνουν αποδεκτοί, αλλά άλλοι χρειάζονται λίγο χτένισμα, πιστεύω. Για παράδειγμα, συμβιβασμό υπαριθμών 1. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τη σωστή, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του σειρά. Καταρχάς ενεργειακή πολιτική και κατά δεύτερον η πολιτική για το κλίμα. Γιατί η πολιτική αυτή θα έχει αποτελέσματα και θα είναι αποδοτική και αποτελεσματική μόνον εφόσον υπάρχει συνολική προσέγγιση και όχι τοπική προσέγγιση. Κατά δεύτερον, πρότεινα να εστιαστούμε στην ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη και όχι τόσο στις παγκόσμιες προκλήσεις. Οι παγκόσμιες προκλήσεις δεν έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, εδώ σε αυτές τις τροπολογίες θα ήθελα να αλλάξουμε την ε, διατύπωση όπου αναφέρεται ότι η αποδοτικότητα της ενεργειακής κατανάλωσης αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για να πετύχουμε την ανεξαρτησία από την εισαγόμενη ενέργεια. Πρόκειται για ένα μόνο εργαλείο Ανθρωπολογία 2. Να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η ενέργεια για την ανταγωνιστικότητα της ενεργειάς μας, για την οικονομία μας. Αν ε, η βιομηχανία μας ε, δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ενέργεια, δεν πρόκειται να είμαστε ανεξάρτητοι. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να διαγράψουμε τις αναφορές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες ή να εφαρμοστούν αυτά παντού. Γιατί θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και ομοιογένεια στη διατύπωση. Αν λοιπόν σε κάποια σημεία, σε τροπολογίες αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία, ενώ σε άλλα σημεία δεν αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία, δεν υπάρχει συνοχή στο κείμενο. Τροπολογία υπαρτιμών 3. Νομίζω ότι αν θέλουμε να θέσουν το θέμα των άμεσων άλλων ε, επενδύσεων, θα πρέπει να γίνεται ε, αναφορά στις υποδομές ε, μεταφοράς, όχι οποιασδήποτε υποδομές, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Να φανταστούμε να μην επιτρέπονται οι αλλαδοτές άμεσες επενδύσεις στην Ευρώπη σε θέματα ενέργειας. Παλιά είχαμε μόνο τις εθνικές ε, εταιρείε. Αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Και πιστεύω επίσης ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αναφέρεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενέργεια και όχι μόνο σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και της σχετικής νομοθεσίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτελεί όμως ένα μόνο το μήμα του συνόλου. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό μόνο. Επίσης να διαγραφεί η αναφορά στο, στην ισοτιμία ε, ευρώ-δολαρίου. Καταλαβαίνω ποια είναι το σκεπτικό, αλλά πιστεύω ότι δεν ταιριάζει εδώ αυτή η αναφορά. Η τροπολογία 4 και η τροπολογία 5 μας βρίσκουν σύμφωνους, ή συγγνώμη, λύσει, λύσεις, συμβαστικές τροπολογίες 4 και 5. Στη συμβαστική 6 θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στην ευρωπαϊκή και πάλι διάσταση και όχι στις παγκόσμιες ε, προκλήσεις και να διαγραφεί η φράση ενεργειακή αποδοτικότητα παγκοσμίω. Μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το υπενθυμίζω. Ακόμα και αν ε, υπάρξουν ε, εξελίξεις ας πούμε, στην Αφρική ή στην Ασία, δεν θα μας βελτιώσει αυτή την ενεργειακή ασφαλεία στην Ευρώπη. Στο σημείο μόνο 7, στο συμβαστική τροπολογία 7. Πιστεύω ότι είναι πολύ περιορισμένη η αναφορά στην ενεργειακή αποθήκευση και στην ε, πράσινη ενέργεια. Συμφωνώ μεν αλλά αν κάνουμε τέτοιο περιορισμό στο έγγραφο αυτό που αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, αν είναι τόσο περιορισμένο το πεδίο μας, δεν θα καταφέρουμε όσα θα έπρεπε. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε μόνο στην ενεργειακή αποθήκευση και μετά να περιορίσουμε αυτόματα και το είδος της ενέργεια που θα πρέπει να αποθηκεύεται. Και επίση είναι περιττό να γίνεται αυτός ο να γίνεται αυτή η αναφορά στην ανάγκη κατάργησης των μασμολογικών φραγμών. Οι τεχνολογίες που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποδομές. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιασδήποτε τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την ανεξαρτησία και την ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ευρώπη. Αυτό θα ωφεληθεί και εμάς και τις τρίτες χώρες, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κυρία Σέινφελτ, για τους ε, σοσιαλδημοκράτες ε, εισηγητής είμαι εγώ και θα πάρω λοιπόν το λόγο ως ε, σκιώδη. Κύριε Σέινφελτ, όντως πιστεύω ότι το θέμα της παραγωγής ενέργειας σε άλλες χώρες, σε, σε τρίτες χώρες, έχει να κάνει και με τη δική μας ενεργειακή ασφάλεια. Αν η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται για πρώτες ύλες, θα είναι διαφορετική κατάσταση στον ανταγωνισμό. Θα μας επηρεάσει αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν το θέμα των τρίτων χωρών είναι σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια και ο προσανατολισμός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί ένα τρόπο για την σταθεροποίηση της ενεργειακής προμήθειας. Ιδιαίτερα εφόσον σε τρίτες ε, χώρες χρησιμοποιούνται ε, τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και ενεργειακές πήγες ε, από τις οποίες αφαιρείται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Έχουμε μέχρι το 50% στην παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τις εμπορικές συμφωνίες. Η διάσταση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτές τις ε, διμερείς συμφωνίες. Και τρία σημεία με απασχολούν ιδιαίτερα τα οποία αποτυπώνονται και στις συμβαστικές τροπολογίες. Αφενός, να διατυπώσουμε ασφαλώς σε εμπορικές συμφωνίες ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται για dumping σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας. Γιατί αυτό φυσικά διαμορφώνει διαφορετικές μορφές εξάρτησης και δομές εξάρτησης. προκειμένου επιτέλου να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα τη ε, ζήτηση και της μείωσης της ζήτησης. Ε, κατά δεύτερον, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εμπορικές συμφωνίες όπου θα εισαχθούν σχετικά α, κεφάλαια για την ενέργεια. Αυτό το συζητάμε σε διάφορες διμερείς ε, συμφωνίες και σε ό,τι αφορά το θέμα του προσανατολισμού της ενεργειακής πολιτικής και το θέμα της ε, διαφοροποίησης των σχετικών υποδομών παραγωγής ενέργειας, το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας. Για όλα αυτά τα θέματα λοιπόν αξίζει τον κόπο να κάνουμε συμφωνίες σε ό,τι αφορά διμερείς ε, ε, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες και να συμφωνήσουμε επί προτύπων ποιότητας προκειμένου το θέμα της ενέργειας να ενταχθεί πιο βιώσιμα στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και να μην ε, υπονομεύεται. Και θα ήθελα αυτό το σημείο να συμπεριληφθεί γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό και για την Επιτροπή Εμπορίου. Είναι καθοριστική σημασία στο σημείο αυτό. Τρίτο στοιχείο που με απασχολεί, το θέμα των ενεργειακών συμβάσεων με τρίτες χώρες. Και εδώ όντω. πριν από κάποια χρόνια είχαμε κάποια νομοθεσία, αναπτύξαμε νομοθεσία για μεγαλύτερο συντονισμό της ενεργειακής πολιτικής με τέτοιες χώρες. Αλλά το Συμβούλιο των Υπουργών αρνήθηκε να εγκρίνει την νομοθεσία αυτή προέκυψε μια υποχρέωση ενημέρωση των κρατών μελών προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό δεν σημαίνει συντονισμό τη ενεργειακή πολιτική με τρίτα κράτη. Ο Helmut Σόλτ επισήμανε ότι συζητάμε εδώ και πολύ καιρό την έκθεση αυτή και εδώ και κάποιες εβδομάδες βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση όπου εκ νέου ανοίγει το θέμα αυτό και δικαίω στην νομοθεσία που έχουμε μπροστά μα περιλαμβάνεται και μια ρετρένα θεώρηση. και εγώ θεωρώ ότι μάλλον είναι αυτονόητο ότι θα μα κάνει κάποια πρόταση αναθεώρησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί, θεωρώ, είναι ότι σε ένα τέτοιο πακέτο ενεργειακής ε, σύμβασης, ε, ενεργειακών συμβάσεων ε, με τρίτες χώρες, να υπάρχει μια εξάντε αξιολόγηση. Και ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και στην ιστορική αγορά της ενέργειας. Αλλά αυτό που είναι απαραίτητο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την κατάρτιση συμφωνιών με τρίτες χώρες να συμμετέχει για να υπάρχει συντονισμένη στρατηγική. Και τέλος, διαπιστώνουμε συνέχεια ότι το θέμα των ενεργειακών συμφωνιών και της σχετικής ενεργειακής στρατηγικής είναι κάτι το, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα τρία στοιχεία λοιπόν θα ήθελα να συμπεριληφθούν στην έκθεση. αλλά διαπιστώνω ότι έτσι κι αλλιώ προ την κατεύθυνση αυτή αναπτύσσεται και προσανατολίζονται οι συμβιβαστικέ τροπολογίε. Ο κύριο Σαράλντι είναι υπεύθυνο από το ECR, αλλά θα πάρει το λόγο η ΕΜΑ. Ευχαριστώ. Δυστυχώ ο σκιώδη μα Ζαχαράντιλ δεν είναι παρόν. Τον εκπροσωπώ. Καλωσορίζει την εργασία του εισηγητή και την πρώτη προσπάθεια συμβαστικών τροπολογιών. Καλή για συζήτηση καλωσορίζει το γεγονός ότι πολλά στοιχεία των τροπολογιών της ομάδας μας λύθηκαν υπόψη, αλλά πρέπει να κάνουμε περαιτέρω προσπάθειες για να είναι κοινώ αποδεκτή η προσπάθεια συμβασμών. Έχουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πολλές τροπολογίες ασχολούνται με εσωτερικά θέματα της Ένωσης. Αυτό είναι θέμα ήτρε η ίντα πρέπει να ασχοληθεί με τις δικές της αρμοδιότητες, να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην επί της ε, αρμόδια επιτροπή για τη σημασία του θέματος αυτού. Έχουμε κάποια προβλήματα για αυτά που λέγονται για, τον, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα όπου η Επιτροπή και πολλές ομάδες εξέφρασαν πολλές ανησυχίες για το τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού μηχανισμός για το εμπόριο δικαιωμάτων παγκόσμια για το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν θέλουμε να ξαναρχίσει η συζήτηση για τα, τις αμυντικές ε, συμφωνίες. Να μην ξαναρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Ανησυχούμε επίσης για τις τροπολογίες που ασχολούνται με συλλογικές συμβάσεις αγορών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν πώς συνεργάζονται για κοινή αγορά ενεργειακών προϊόντων. Μπορεί να θεωρείται ελκυστική από κάποιους, αλλά το βασικό μήνυμα πρέπει να είναι ότι η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει την εμπορική πολιτική για να διαφοροποιήσει τις ε, ενεργειακές της προμήθειες παντού στον κόσμο για να μην εξαρτώμεθα από ένα σημείο αγοράς και μεταφοράς. Αυτό είναι το θέμα. Ο κύριος Ζαχαραντήλ, ευχαριστή και πάλι τον εισηγητή καλωσορίζει την εργασία του για αυτήν την σημαντική ε, και σκόπιμη σε αυτή τη φάση προσπάθεια. Ευχαριστώ οι φιλελεύθεροι δεν είναι παρόντες, λέει ο Πρόεδρος, για τους πρασίνους. Ισκά Ευχαριστώ. Από πλευρά του δικού μου σκιώδου, Μπούχνερ, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Στο συνάδελφο από το ΕΛΚ να πω ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση λοιπόν ε, της κατοικησιμότητας του πλανήτη δεν ξέρω αν είναι τόσο δευτερεύον θέμα. Όλοι πρέπει να επιλύσουμε αυτό το σφαιρικό πρόβλημα. Αν πούμε απλώς ας αφήσουμε όλες τις ζητήσεις σε σφαιρικό επίπεδο να ασχοληθούν με αυτό δεν θα κάνουμε τίποτα. Η βιωσιμότητα, το περιβάλλον πρέπει να είναι τμήματα οποιασδήποτε στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Γιατί και αυτό ασφάλεια είναι για το μέλλον. Ας δούμε τι γίνεται στο Βανουάτου για να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το θέμα αυτό. Ο Σκιώδης μας συμφωνεί με τον εισηγητή ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την αύξηση αποδοτικότητας, της νέες τεχνολογίες, τις εναλλακτικέ ενέργειες και τη μείωση της οικιακής κατανάλωσης. Κάποιες διατυπώσεις που έχουμε προτείνει στις τροπολογίες μας θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις συμβαστικές που έχουν προταθεί, για παράδειγμα στην 7 που ασχολείται με την αυξανόμενη χρηματοδότηση της αποθήκευσης της ενέργειας, να βάλουμε αυτά που λέμε ότι η τεχνολογία για την αποθήκευση και την μεταφορά από ανανεώσιμες μετατρέποντάς την αυτή την ενέργεια σε φυσικό αέριο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί εδώ. Επίσης, διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας πρέπει να συμβαδίζει με τις εσωτερικές μας πολιτικές. Να μην ανοίξουμε δηλαδή τώρα την πόρτα στην υδρορογμάτωση ε, και τις ε, σχιστολιθικές άμμους. Και πάλι λοιπόν ευχαριστώ τον εισηγητή και ο σκιώδης μας ε, ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Α, οπότε ο Βίκτορ μετά. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτζε για την ε, τόσο αποδοτική συνεργασία που είχαμε. Πάντα ήταν διαθέσιμος και επίσης θα πρέπει να του πω ότι του υπόσχομαι τελικά να έχουμε τέτοιες συμβασκετοπολογίες που να ε, αντικατοπτρίζουν όλες τις τάσεις και ακριβώς όπως ε, θέλουμε ως Επιτροπή να είναι τα πράγματα γιατί ακριβώς εδώ το διεθνές εμπόριο ε, γίνεται πράξη μέσω των συνθήκων και μέσω της πολιτικής που ασκούμε ενέργεια, ενεργειακή ασφάλεια κλπ. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες που να έχουν και αυτή, την, πλευρά την ενεργειακή. Επίσης τώρα μιλούμε για ενεργειακή ασφάλεια με δύο διαστάσεις. Πρώτα πρώτα την ασφάλεια προσφοράς και παροχής, κάτι το οποίο έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Σήμερα με την κρίση στην Ουκρανία και επίσης με τη σχέση Ουκρανίας-Ρωσίας γενικότερα. Ε, επίσης από την άλλη μεριά έχουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος του ενεργειακού ή στην ασφάλεια του κάθε κράτους. Μα σήμερα ενέργεια σημαίνει ασφάλεια. Ρίξα μια ματιά στις εξελίξεις. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι ε, στην παγκόσμια σκηνή η ενέργεια έχει σημαινει ασφαλεια ριξε μια πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Ακριβώς όπως είπαμε για ε, την Ουκρανική κρίση, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και θέματα ενεργειακά Έχουμε αυτή τη συμφωνία 400 δις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Και εντάξει, αυτά είναι νούμερα. Αλλά πρόσφατα διάβασα ότι ίσως η Κίνα μπορέσει να αποκτήσει 50, 50 σημεία εξόριξης, άντλησης τέλο πάντων φυσικού αερίου στη Ρωσία. Ακριβώς γιατί υπάρχουν προβλήματα της παροχέτευσης του αερίου από τη Ρωσία. Επίσης, για, το, για την υδρορογμάτωση. Όσον αφορά τη ΣΥΠΑ είδατε τι μειώσεις επιφανειακές είχαμε για το αέριο που παράγεται έτσι. Είδατε τι να συνέβη στη διεθνή αγορά. Επομένως, θα πρέπει να τονίσουμε το ότι χρειάζεται μία προσπάθεια συντονισμού που να είναι συστηματική. Να συνδυάσουμε τις εμπορικές συμφωνίες με την ε, πολιτική ασφάλειας αλλά και την εξωτερική μας πολιτική. Αυτό το πρεσβεύει η πολιτική μας ομάδα, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό έχουν δεσμευτεί οι επίτροποι, τα είπαν αυτά τότε στις ακροάσεις τους, άρα να είμαστε συνεπείς με τα όσα υποσχεθήκαμε. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι διατυπώσεις που έχουμε όπως ε, εναλλακτικέ πηγές, ε, κλπ. Να γίνονται πράξη, όχι μόνο να τα λέμε, αλλά να τα εντάσσουμε αυτά στις εμπορικές συμφωνίες, τόσο ώστε αυτές οι εναλλακτικέ ε, πηγές προμήθειας να αποτελούν μια πραγματικότητα και έτσι να έχουμε λιγότερη εξάρτηση από τον ένα προμηθευτή. Να το σημερινό πρόβλημα. Επίσης, το ίδιο σημαντικό είναι και κάτι άλλο να δούμε πώς στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες θα έχουμε ένα κεφάλαιο που να αφορά την ενέργεια. Ακριβώς πώς κανουμε και στο TTIP. Και έτσι τα πράγματα να είναι προβλέψιμα. Να δει από κάποια σταθερότητα οι μελλοντικέ εξελίξεις και όσον αφορά το κεφάλαιο ενέργεια. Εν κατακλείδη θέλω να σας πω για τις ε, διαπραγματεύσεις με τρίτους. Ωραία να τονίζουμε τον ρόλο των κρατών μελών. Ή να λέμε για αυτούς οι οποίοι εκούσια ε, και με ητοπάθεια πάνε να μιλήσουν στην Κασπρόμ. Όμως, για φανταστείτε, ε, τα κράτη-μέλη που έχουν σημαντικά προβλήματα, εάν κάτσουν να διαπραγματευτούν με κάποιον ισχυρό συνομιλητή, τότε πώς θα πετύχουν κάτι καλό για τον εαυτό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που είπε ο Μάρος Σεύκοβιτ, δηλαδή να γίνεται η διαπραγμάτευση μόνο στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να έχουμε γενική εφαρμογή της ενεργικής πολιτικής μας. Ξανά να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σόλτς για το πόσο διαθέσιμο ήταν για την ε, προθυμία του και για το ότι μου υποσχέθηκε τέσσερα τροπολογίες μου πρόκειται να ενταχθούν στο κείμενο στις ε, συμβασιές τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα είμαστε στο περιστάσιο μας αφορά την, την καινούργια εποχή στην ενεργειακή πολιτική. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Um, Σα ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και για την ποιότητα τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή που εστιάζεται τέτοια πολύ στην πτυχή του διεθνού εμπορίου. Θα θέλαμε εδώ να τονίσουμε τη σημασία τη εξωτερική διάστασης στην Ενεργειακή Ένωση που πρόσφατα εγκρίθηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται για μία από τις ε, πέντε πτυχές της ενεργειακής ε, ασφάλειας και της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι σαφές ότι το διεθνές εμπόριο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για να ε, μπορέσουμε να αγγιηθούμε την ενεργειακή ασφάλεια. Να περάσουμε λίγο στις λεπτομέρειες τώρα της διάστασης της Ενεργειακής Ένωσης και σε ό,τι αφορά την εξωτερική πτυχή βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι γεωγραφικοί τομείς που έχουν υπογραμμιστεί. Η ιδέα ενίσχυσης ενεργειακών εταιρικών σχέσεων με βασικούς εταίρους όπως η ΕΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία. Φυσικά το εμπόριο θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διδραματίσει για την ανάπτυξη μια συνεκτικής στρατηγικής LNG σε ό,τι αφορά το θέμα της εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η δεύτερη ιδέα είναι η στρατηγική σχέση με βασικές χώρες παραγωγής όπως η Τουρκία, το, η Αλγερία, το Αζερβαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν αλλά και αφρικανικές χώρες. Και εδώ πάλι η πτυχή του εμπορίου στις στρατηγικές αυτές εταιρικέ σχέσεις θα είναι ουσιώδης. Τέλος, θα ήθελα μεταξύ άλλων να αναφέρω δύο γεωγραφικές ε, περιοχές. Θέλουμε να αναπτύξουμε το πλήρες δυναμικό των χωρών της ε, Μεσογείου για να αναπτύξουν τις υποδομές για το υγροποιημένο αέριο, αλλά και για, και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στην Κασπία θάλασσα, όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και αερίου. Επειδή λοιπόν είναι τόσο σημαντικές αυτές οι γεωγραφικές περιοχές, φυσικά οι εμπορικές σχέσεις θα έχουν μεγάλη σημασία για τη διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις περιοχές αυτές και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, τα ενεργειακά κεφάλαια στις εμπορικές ε, συμφωνίες, αλλά και σε ό,τι αφορά τη μορφή των συμφωνιών αυτών. Το θέμα λοιπόν των συγκεκριμένων, της που θα πρέπει να εισαχθεί σε κάθε περίπτωση στις συμφωνίες, για παράδειγμα ρήτρες προορισμού, προκειμένου το αέριο που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κυκλοφορεί μετά ελεύθερα στην αγορά. Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί πρόβλημα. Και αυτό αποτυπώνεται και στις σχετικές διακυβερνητικές συμφωνίες που συνήθισαν πριν από κάποια χρόνια Τέλο να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώ παραμένει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. σα ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ την Επιτροπή σα και το σύνολο του Κοινοβουλίου για την μεγάλη πολιτική δέσμευση για θέματα ενεργειακή ασφάλεια και ασφαλώ αυτό έχει βοηθήσει στο να τοποθετηθεί στο επίκεντρο τη Ενεργειακή Ένωση, η Ενεργειακή Ασφάλεια. Και θέλουμε λοιπόν να συγχρονιστεί και αυτή η άσκηση με το ζήτημα της εφαρμογής της Ενεργειακής Ένωσης και στα διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Χέλμου, θες να σχολιάσεις. Δεν θέλω να με ακρηγορήσω, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και τους κοιόντες και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, υποστήριξή της. Τρία σημεία. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια τη συζήτηση προέκυψε σαφώ ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο ένα ιστορικό ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι 28 χώρε, αλλά έχει και μια παγκόσμια διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τα συμφέροντα και τη σημερινή αλλά και τη μελλοντική γενιά ε, θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή ενέργεια, σε επαρκή ενέργεια για να μην υπάρξει ενεργειακή φτώχεια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει με το πώς ε, συμπεριφέρεται η Ευρώπη των 28 σε σχέση με τις άλλες χώρες, πώς συνεργάζεται για την κοινή ενεργειακή παροχή και παραγωγή. Να μην ξεχνάμε λοιπόν αυτή την παγκόσμια διάσταση. από πλευρά τη οικονομική κατάσταση των κρατών μελών. Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. το λύθιο, σε ό,τι αφορά το λύθιο, πολλοί για τον τομέα της ε, παραγωγής ενέργεια μα λένε ότι μετά το πετρέλαιο θα έρθει το λύθιο. Σε συνδυασμό με τον άνθρακα έχουμε ανθρακούχο λύθιο. Αυτό τι σημαίνει ότι αν σκεφ... θέλουμε να σκεφτούμε θέματα αποθήκευσης θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πού είναι τα μισά αποθέματα της ε, παραγωγής ε, του λιθίου στη Βολιβία. 13 εκατομμύρια τόνοι. Μεγάλη ποσότητα, μεγάλος όγκος. Πώς λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ πηγές ενέργειας, θα πρέπει να έχουμε μοντέλα συνεργασίας. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για νέα μοντέλα Ενεργειακή αποδοτικότητα. Ήδη από σήμερα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα τη ενεργειακή ασφάλεια και τη ενεργειακή ε, της ασφάλειας ενεργειακής παροχής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και εδώ να προωθήσουμε και την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να ενταχθεί στις εμπορικές συναλλαγές και με τις τρίτες χώρες. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπάρξει σαφής περιχαράκωση. Προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε με τις συμβαστικές τροπολογίες προκειμένου να είναι λογική η χρηματοδότησή μας και να εξυπηρετεί τους σκοπούς μας τους σκοπούς της ενεργειακής ασφάλειας και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή σε μια ενεργειακή ένωση. Δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να αναφέρω. Ε, επειδή το έθεσε και ο συνάδελφος Μπαστινάρου. αν είχαμε σκεφτεί ήδη εγκαίρως ε, πώς στη Ρωσική Ομοσπονδία μπορούσαμε να ξεχρονίσουμε την παραγωγή της ενέργειας, ίσως θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε λιγότερα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Να αναφέρω μία διάσταση για την οποία θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε. Και θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι και άλλες χώρες με τις οποίες ε, έχουμε εμπορικές συμφωνίες, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ενεργειακό κεφάλαιο και να οριστεί με σαφήνεια το θέμα της ε, ενεργειακής ασφάλειας αλλά και της βιωσιμότητας. Στη διάσταση λοιπόν αυτή θα πρέπει να κάνουμε υποχώρηση και προς τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί και αυτοί θα πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα αποφύγουν την ενεργειακή φτώχεια. Αυτό φυσικά αφορά και την Αφρική και την Εθνική Αμερική, την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Ως εκ τούτου. Θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια εδώ πόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα προς το συμφέρον όλων τελικά σε ό,τι αφορά και τους ε, αναπτυξιακούς στόχους. Και τέλος. Προσπαθώ να συμπεριλάβω τα σχόλια που άκουσα, ακόμα και αυτά που ίσως είναι λίγο πιο επικρατικά, για να είμαστε επικοδομητικοί τελικά. Ωραία, θα ψηφίσουμε στις 14 Απριλίου. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 14. Το νομοθέτημα για τα λεγόμενα κορυφτά συγκρούσεων έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες μας και πώς μπορούμε να τις προμηθευόμεθα υπό ε, σωστές συνθήκες. Ο κύριος Βέγκλερ είναι εισηγητής μας. Για την έκθεσή του έχουν υποβληθεί εδώ μεταξύ 576 τροπολογίες. για τις οποίες θέλουμε να ψηφίσουμε τον επόμενο μήνα. Πρέπει λοιπόν κάπως να διευκρινίσουμε την κατάσταση, να δούμε σε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οι δύο επιτροπές που έπρεπε να μας δώσουν γνωμοδοτήσεις ε, ψήφισαν. Η ΝΤΕΒΕ μας έστειλε μία γνωμοδότηση με 50 τροπολογίες. Είναι αρκετά ομοιογενής. Η ΑΦΕ δεν έχει κάνει γνωμοδότηση ακόμη, δεν τα έχει καταφέρει. Γιατί κατά την τελική ψηφοφορία ισοψήφισαν υπέρ και κατά, 12 υπέρ, 12 κατά και 43 αποχές. Οπότε δεν εγκρίθηκε η έκθεση. Οπότε δεν έχουμε τροπολογίες. Από την Άφετ μόνο λίγες από την ΤΕΒΕ. Κύριε Βίγκλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, αν είχαμε γνωμοδότηση από την ΑΦΕΤ θα είχαμε άλλες 50 από ό,τι φαίνεται τροπολογίες. Πολύ σωστά περιγράψατε την κατάσταση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους Κιώδης και όλους ε, που με βοήθησαν από τις πολιτικές ομάδες για να εκπονήσουμε αυτό το πολύ περίπλοκο κείμενο. Ευχαριστώ και δημοσίως, ε, θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή συνεργασία. Το συζητήσαμε επανειλημμένα. Ευχαριστώ επίσης για την πολλή εργασία που έχει κάνει και αυτή που θα κάνει ακόμη η γραμματεία μας. Είναι νομίζω σαφές, σαφέστατο, ότι έχουμε καθυστερήσει. Χρειαστήκαμε έναν επιπλέον μήνα, αλλά έχει συμφωνηθεί αυτό μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τον ε, πολύ μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Και ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να είναι λειτουργικός, να επιτύχει το στόχο του. Λοιπόν, ο εμπορικός κανονισμός που συζητάμε είναι ένα στοιχείο της λεγόμενης ολοκληρωμένης ενωσιακής προσέγγισης, η οποία προσέγγιση βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ένας από τους πυλώνες είναι αυτός ο οργανισμός για το σύστημα αυτοπιστοποίησης, για τη δέωση επιμέλεια, για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των ορυκτών. Ο δεύτερος πυλώνας που αναφέρει η συνοδευτική ανακοίνωση που είναι κοινή μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής και του προσώπου είναι τα συνοδευτικά μέτρα για να βοηθήσουμε τις εταιρείε της Ένωσης για να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα αυτοπιστοποίησης και ο τρίτος πυλώνας είναι τα συνοδευτικά μέτρα που θα εφαρμόσουμε μέσω πολιτικών, διπλωματικών και αναπτυξιακών ενεργειών συνεργασίας επί τόπου στις περιοχές όπου υπάρχει υψηλό κίνδυνος ή σύγκρουση. Ως εισηγητής θεωρώ ότι ο κανονισμός πρέπει να πληρεί πολλές προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματικός, να λειτουργεί και να έχει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να λάβει υπόψη την πείρα που έχουμε συλλέξει να συμπεριλάβει τους μηχανισμούς που ήδη λειτουργούν και τις πρωτοβουλίες ε, του κλάδου. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να υπάρξει ουσιώδη συνεργασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμφωνούν. Γιατί παίζουν ρόλο όλοι αυτοί ή μπορεί να παίξουν ρόλο στην αλλαγή της κατάστασης επιτόπου. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Να αλλάξει η κατάσταση. Ναι, μεν αναφερόμεθα στη δημοκρατική δημοκρατία του Κόγκο, αλλά μπορεί να θέλουμε να αναφερθούμε και σε άλλε περιοχέ όπου υπάρχουν συγκρούσει ή υψηλό κίνδυνο σύγκρουση. Και επίση πρέπει να είναι αναλογική αυτή η ρύθμιση. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε μονομερό στι επιχειρήσει μα ε, υποχρεώσει. Πρέπει να είναι επίση όφρονη νομοθεσία. Γιατί αφορά και ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων. Πάντα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα της μικρομεσαίας, Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά <clears throat> της οικονομίας μας. <clears throat> Ο κανονισμός πιστεύω θα έχει μία σαφή ρήτρα αναθεώρησης. Δηλαδή θα εκτιμήσουμε πώς λειτουργεί ο κανονισμός επιτόπου στις περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις και πόσο συμμετέχουν οι εταιρείες από την Ένωση. Και επίσης θέλουμε να δούμε και πώς θα αλλάξουν ενδεχομένω οι καθευτήρες γραμμές ε, της δέουσας προσοχής του ΟΣΑ. Επιπλέον. Να λάβουμε υπόψη ότι οι εμπορικοί κανονισμοί θα πρέπει να παρεμποδίζουν την παρέκκληση του εμπορίου. Δηλαδή να σταματήσει το εμπόριο σε αυτές τις περιοχές και να πάει αλλού. Και επίσης να μην έχουμε τίποτα ανεπιθύμητα ε, αποτελέσματα εμπάργκο. Θέλουμε να υπάρξει ένα λειτουργικό εφαρμοστικό πλαίσιο. Στα πλαίσια αυτά τονίζω ότι πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία όταν εκτιμούμε τα αποτελέσματα του νόμου Dodd-Frank. Γιατί έχουμε διάφορες αναλύσεις οι οποίες ε, απέχουν πολύ η μία από την άλλη με βάση τις πηγές τις οποίες έχουν βασιστεί. Διάφορες πηγές ενημέρωσης, διάφορες απόψεις. Και κάτι ακόμη, συνάδελφοι. Χθες στην Επιτροπή μας, μάλλον η Επιτροπή μας, Ίντα, η Ντέβε και η Άφετ έλαβαν μία επιστολή από την ύπατη εκπρόσωπο αλλά και από τη Σεσίλια Μάστρον, που είναι η Επίτροπος Εμπορίου και από τον Νίμιτσα πως Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αυτοί οι τρεις υπογράφουν την επιστολή περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα συνοδευτικά μέτρα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λέει ότι η νομοθεσία για αυτά τα ορυκτά μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν είναι μια μιας ευρύτερης προσπάθειας να συμβάλλουμε στην καλή διακυβέρνηση. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζει η επιστολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ε, δοθούν κατά την περίοδο 16-20 ακόμη και 20 εκατομμύρια ευρώ για να προωθήσουμε υπεύθυνη εξόριξη στις περιοχές αυτές. Εντός παρενθέσεων, αύξηση περίπου 500% σε αυτό το τομέα. Επιπλέον λέει ότι οι πόροι αυτοί θα δοθούν για να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις και τις περιφερειακές ε, διοικήσεις για να εφαρμόσουν τις οδηγίες του ΟΣΑ, για να δημιουργηθούν πλαίσια δεούσης επιμελίας, για να προωθήσουν τις μικρής κλίμακας εξορρυκτικές προσπάθειες και να εφαρμοστούν αυτά τα πλαίσια λοιπόν σε εθνικό επίπεδο. Και η βοήθεια θα πρέπει να δοθεί και στην κοινωνία των πολιτών και μη κρατικού οργανισμούς για να βοηθηθεί ιδιαίτερα η περιοχή των μεγάλων λιμνών αλλά σύμφωνα με την επιστολή οι πρακτικές ε, ορθής επιμέλειας πρέπει να εφαρμοστούν και στις χώρες ε, διαμετακόμισης ή προορισμού για να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ισχύσουν και σε όλες τις χώρες όπου πηγαίνουν αυτά τα ορυκτά, ιδιαίτερα χώρες της Ασίας. Έχετε στη διάθεσή σα την επιστολή. Αυτά και τώρα θα ακούσω μεγάλη προσοχή αυτά που έχετε να μου πείτε εσείς. Ευχαριστώ κύριε Βίνκλα. Παρακαλώ Μάρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Αρένα. Ευχαριστούμε και εσά, κύριε Βίνκλε. Δεν ήταν απλό το έργο που επιτελέσατε και χρειάστηκε να επιστατεύσετε όλοι σας την ενέργεια και εσείς αλλά και οι σχεδοσυγητές συνεργαστήκαμε επικοδομητικά δεν θα πρέπει να πλουστεύουμε, να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Να είναι η, η εκούσια προσέγγιση ε, παραγωγική και επίσης ε, να μην ε, ξεφεύγουμε σε ιδεολογήματα τα οποία μας στερούν αποτελεσμάτων. Εγώ θα επανέλθω ακριβώς στα επιχειρήματα που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Για να δω τώρα. Ε, αυτό από τη μία το εκούσιο και την άλλη το υποχρεωτικό. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης, της, της προβληματικής αυτής. είναι αυτά που συζητήσαμε ο εισηγητής και εμείς οι σκιώδεις γιατί έχουμε πάρα πολύ θετική αυτή την επιστολή της κ. Μογκερίνη. Η επιστολή αυτή δείχνει ότι θα πρέπει να δούμε ε, τι ισχύει όσον αφορά την ε, προμήθεια αυτών των πόρων. Θα δούμε φυσικά από, πολλά, από πολλές οπτικές γωνίες, εμείς πάντα αυτό πρεσβεύαμε και γι' αυτό και θα δούμε τι γίνεται με την τοπική διακυβέρνηση και ακριβώ ποιοι είναι οι πόροι που θα έπρεπε να επιστρατευτούν για αυτή την τοπική διακυβέρνηση. Θα πρέπει όλα αυτά να τα υποστηρίξουμε Οπότε και η κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική. Επίσης είναι σημαντική ε, αυτό, αυτό το οποίο, ε, αυτή η επιστολή, γιατί ακριβώς ε, έχουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό και θα πρέπει να υπάρξει μια επίπτωση παγκόσμια και όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα το ξαναδούμε αυτό για το θέμα της υποχρεωτικότητας και της εκούσιας εφαρμογής. Έχουμε τώρα έχουμε αυτού, αυτές τις ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι πρόκειται περί πολύ σημαντικού έργου. Έγινε συζήτηση κοινή και τελικά καταλήξαμε σε έναν ε, συμβιβασμό. Άρα και εμείς θα πρέπει εδώ στην Επιτροπή μας να υποστηρίξουμε αυτή τη δουλειά που έγινε αλλά και τους ε, συμβιβασμούς. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε το τι ισχύει σε αυτές τις περιοχές ε, συγκρούσεων. Είναι σημαντικός ο ρόλος μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω των οικονομικών σχέσεων που έχουμε. Αλλά ο στόχος είναι να αλλάξει το τι ισχύει όσον αφορά αυτές τις χώρες προέλευσης, τις χώρες συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Γιατί είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά την προσέγγιση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ιδεολόγημα ενώ μιλούμε για υποχρεωτική εφαρμογή, αυτή η δέουσα επιμέλεια, όπως ορίζεται από τον ε, όσα, στήριζεται στην θεωρία της μόχρευσης των επιχειρήσεων που ελέγχουν την αγορά. Είναι αυτοί που είναι οι μεγάλοι αγοραστές ας πούμε. Τώρα, πόσο μπορούσαμε να επηρεάσουμε αυτού του μεγάλου αγοραστέ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ε, ένα αποτέλεσμα που θα κατακυριαρχήσει σε όλη την αλυσίδα και να ισχύσει ό,τι θέλει όσα. Αλλά να προσοχή να μην έχουμε κάτι αντιπαραγωγικό. Πρώτα-πρώτα, τι γίνεται με τον πρώτο κρίκο τη αλυσίδας γιατί αν δεν υπάρχει μόχλευση εκεί από τους μεγάλους αγοραστές ε, τότε τι γίνεται. Εάν παραμείνουμε σε ρύθμιση εκούσια, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς όπως και εσείς τα υπεραμεινθήκατε. Ε, άρα θα υπάρξουν συνέπειες και γι' αυτό λέμε εμείς ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ρύθμιση και να υπάρχει και υποχρεωτικότητες που να καλύπτει και αυτούς τους μεγάλους αγοραστές. Ε, επίσης, θα, θα ανατραπεί και το κόδωμα των ρυθμίσεων του ΩΣΑ εάν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητες για όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Και, κατά τρίτο λόγο επίσης, θα έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό ο οποίος θα πριτανεύσει στην ιστορική αγορά και έτσι οι προμήθειες θα αρχίσουν να γίνονται εκτός Ευρώπης. Μα κανένας από τους παρόντες συναδέλφους δεν θα ήταν υπέρ μιας τέτοιας λογικής, γιατί η δουλειά μας εδώ δεν είναι να ε, δουλεύουμε έτσι ούτω ώστε να μας οδηγήσουν να πηγαίνουμε στο εξωτερικό να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να παραμείνουν οι δυνατότητες μας, αλλά να τις αναβαθμίσουμε. Άρα αυτή η ρύθμιση υποχρεωτική δεν είναι ένα διαλόγημα. Είναι η αποτελεσματικό σε σχέση με αυτά που θεσπίζει ο ΩΣΑ για την δέουσα επιμέλεια. Τώρα για την επιστολή μου Γερίνη. Είναι 5% της αγοράς τα διηληστήρια τα ευρωπαϊκά. Όμως μιλούμε τώρα για ρύθμιση επί των 19 από τους 340 της παγκόσμιας σκηνής. Και αυτή η 19 εκουσίως ήδη έχουν ασπαστεί την δέουσα επιμέλεια για την βιομηχανία. Άρα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εσείς υποστηρίζετε είναι μια πρόταση η οποία δεν θα αλλάξει τίποτα. Άρα, τι μας λέει η κυρία Μογκερίνη. Ας αποδεχθούμε αυτό το οποίο συμβαίνει χωρίς να το αλλάξουμε καθόλου. Όμως, για την υποχρεωτικότητα και την αποσματικότητα, εμείς τι σας λέμε ότι θα πρέπει κάτι να κάνει για του 340 τη διεθνού σκηνή, ούτω ώστε εκεί να δουλέψει η μόχλη. Σα το λέει αυτό μια σοσιαλίστρια. Σα μιλά μια σοσιαλίστρια για μόχλευση στην αγορά. Και αυτό θα είναι κάτι που θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα τώρα. Όσον αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, κάτι το οποίο μα απασχολεί όλου. Και ακριβώ εάν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, αυτό θα θίξει. Θα κάνει πιο ευάλωτε τι ΜΜΕ και έτσι θα κάνει πιο βαριά, πιο δύσκολη τη διαδικασία για αυτές. Όταν υπάρχει υποχρεωτικότητα, τότε συμμορφώνεται και η βιομηχανία γιατί είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί. Και το ίδιο ισχύει για όλου του κλάδου, όλου του τομεί παγκοσμίω, γιατί υποχρεωτικότητα αυτό θα πει. Οπότε έτσι διευκολύνονται και οι ΜΜΕ. Γιατί η βιομηχανία δουλεύει επωφελία των ΜΜΕ. Όταν δεν υπάρχει όμως υποχρεωτικότητες τότε έχει τις ίδιες υποχρεώσει με ΜΜΕ, όπω έχει και μια μεγάλη βιομηχανία για να μπορέσει να καλυφθεί, να μπορέσει τόσο να προσχωρήσει στην due diligence. Οπότε είπαμε ότι η μία ρύθμιση θα ωφελεί τι ΜΜΕ, ενώ η άλλη θα αποτελέσει ράπισμα. Θα πρέπει μόνο στους ΜΜΕ να δουν τι θα κάνουν, κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο, κάτι το οποίο θα είναι δαπανηρό. Άρα πάνε ΜΜΕ. Οπότε για άλλη μια φορά σας λέω ότι, θα, ότι είναι λάθο να λέμε ότι η υποχρεωτικότητα είναι ιδεαλισμός ή κλπ. Το αντίθετο ισχύει. Ιδίω για τις ΜΜΕ. Γι' αυτό σα λέω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και τα έχουμε πει με όλου τους εμπλεκόμενου σε όλη τη διαδρομή της ε, αλυσίδα παραγωγής. Μη και οργανώσεις, εκπρόσωποι του Business Europe, Μιλήσαμε με όλους, όλους. Και τα επιχειρηματά τους είναι βάσιμα. Άρα κλείσουμε ένα συμβασμό, το ώστε τελικά να έχουμε μια ρύθμιση αποτελεσματική. Γιατί, κύριε Σιγητά, αυτό θέλουμε, αποτελεσματικότητα. Ο πρόεδρος. Uh, uh, Ευχαριστώ, έμα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ξεκινήσει ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή για το έργο που έχει κάνει και για την συνεδρίαση των σκιωδών την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ακόμα και αν ε, δίστανται οι απόψει μεταξύ των ομάδων για το πώ φανταζόμαστε εμεί ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη εξόρεξη κάποιων ορεικτών και της, ε, των συγκρούσεων στι περιοχέ αυτέ. Όλοι θέλουμε ασφαλώ να λυθεί το πρόβλημα αυτό με τον όποιον τρόπο. Υποστηρίζουμε γενικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε καταθέσει πιο λίγες τροπολογίες από πλευρά του ECR για να διευκρινίσουμε κάποια από τα στοιχεία τα οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση. Θέλουμε η διατύπωση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι ρεαλιστική. Άρα αν λέμε self-declare αντί για self-certify, θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σωστό. Όταν δηλαδή δηλώνουμε ότι εμείς εφαρμόζουμε δέουσα επιμέλεια, η διατύπωση είναι πιο σωστή. Επίσης, ε, να γίνεται αναφορά σε περιφερειές και όχι σε περιοχές. Πολύ απλά για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνοχή μέσα στο κείμενο. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, ωστόσο, το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε εμείς ως βουλευτές, είναι ότι η βιομηχανία σε κάποιο βαθμό ήδη εφαρμόζει κάποιες δικασίες δέουσας επιμέλειας. Και κατανοούμε ασφαλώς ότι οι καταναλωτές είναι όλο και πιο απαιτητικοί για τα προϊόντα που αγοράζουν. Θέλουν να μην προέρχονται από εμπόλεμες καταστάσεις, όπως το πρόγραμμα το οποίο εγγυάται ε, ότι δεν προαγάγονται οι συγκρούσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε ενδεχόμενες αλληλεπικαλύψεις για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα τα οποία θέλουμε και να αναγνωρίσουμε επαρκώς τα πρότυπα αυτά. Κάτι το οποίο επεσήμενα στη συνεδρίαση των σκιωδών και στις συζητήσεις που έχουν λάβει η χώρα εδώ στην Επιτροπή είναι το γεγονός ότι όλες οι ομάδες λαμβάνουν υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και μπορεί η ιδέουσα επιμέλεια να είναι κάτι σχετικά απλό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεγάλους ομίλους. Μπορεί να είναι μεγάλη η διαφορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό λοιπόν με απασχολεί ο αντίκτυπος αυτές τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στη δική μου περιφέρεια ο αντίκτυπος που θα υπάρξει στις μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον ενδεχόμενο αντίκτυπο και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο το οποίο θα εξηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπει ο κανονισμός. Θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικά κρίσιμος πόρος αυτός για όλες τις επιχειρήσεις, οποιαδήποτε μεγέθους. Ιδιαίτερος ε, επειδή ο κατάλογος ε, των εμπόλεμων περιοχών δεν θα περιληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να αγγιηθούμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Έχουμε επίση τροποποιήσει την ιδεολογική σκέψη παριθμών 12 που παρακολουθεί τον αντίκτυπο του κανονισμού και προτείνει έλεγχο από τρίτη μέρη, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό αυτό, θέλουμε πραγματικά να γνωρίζουμε το κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις μας, ε, γιατί είναι κρίσιμες για την οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν τον αντίκτυπο της ε, νομοθεσία. Και νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε, μια γενικότερη, σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναγκών, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ωστόσο το πλαίσιο αυτό, προκειμένου να είναι πιο σταθερή, πιο τακτική η έλεγχη κάθε τρία χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. εκτιμώντα τον αντίκτυπο της νομοθεσίας, οποιοδήποτε μηχανισμό, επιτόπου, στους τομείς αυτού. Υπάρχει διαφορά, επηρεάζεται, το πρόβλημα απαλύνεται, αμβλύνεται. Είναι ουσιώδος σημασία σε αυτό. Και όποια προσέγγιση και να ακολουθήσουμε, η νομοθεσία θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς, προκειμένου να προσαρμόζεται ανάλογα με τι εξελίξει και για να δούμε τι έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, διέλαβα ότι στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Δεν θέλω η νομοθεσία να έχει αρνητικό αντίκτυπο βάσει με μια αξιολόγηση που έγινε από τον Φρανκ. Θα πρέπει πλήρως να κατανοήσουμε τον ακριβή αντίκτυπο παντού εδώ λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθεί το έργο μα. Και αυτό θέλω να κάνω και σκοπεύω να κάνω με τους συναδέλφου μου τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρος. Έλμουτα, έχετε σκιώδη. Α, εσύ είσαι σκιώδη. Ähm, και εγώ ευχαριστώ. Τον Σαλφο Βίγκλα για τη συνεργασία που είχαμε για αυτό το σημαντικό τομέα. Βδομάδες τώρα συνεργαζόμεθα. Παρά το ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις ή θέλουμε να τονίσουμε διαφορετικά θέματα. Ορισμένα υπόθηκαν κατά την τρέχουσα συζήτηση. Να πω ευθύ εξ αρχής ότι κάναμε και μια κρόαση για το θέμα αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αναγκαιότητα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος. Γιατί εμείς ως Ένωση γιατί να μην συμφωνήσουμε, γιατί να μην συμφωνήσουμε με τις κατευθύνες γραμμές του ΩΣΑ που λένε για μια σωστή και διαφανή εφαρμογή πολλά θέματα, το θέμα της ε, δεσμευτικότητας. Πολλά θέματα τα έχουν ήδη εφαρμόσει τα κράτη-μέλη. Τονίστηκε η σημασία του και η αναγκαιότητα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι να επιδείξουμε συνέπεια με τη στάση μας εντός του ΟΣΑ. Διότι ως κράτη-μέλη του ΟΣΑ έχουμε αποφασίσει αυτές τις κατευθυντήρες, γιατί λοιπόν να μην τις συμπεριλάβουμε τώρα στη δική μας νομοθεσία, όπως είπε η Αλφουσα Αρένα. Και εδώ υπάρχει η βασική διχογνωμία μεταξύ των ομάδων, αν θα πρέπει να είναι εθελουσία η συμμετοχή ή υποχρεωτική αυτή η οδηγία. Όλα όσα συζητήσαμε με τους εκπροσώπους του ΟΣΑ, με εκπροσώπους από τις ε, μεγάλες λίμνες, όλοι μας είπαν ότι θέλουν να λάβει σαφή θέση της Ένωσης, άρα και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που είναι οι συνομοθέτες. Πρέπει λοιπόν να τολμήσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα. Και υπάρχει και το βραβείο Ζαχάροφ το οποίο έχουμε δώσει και αυτό μας είπε ο εκπρόσωπο, ο, αυτό μας είπε ο διακεκριμένος κάτοχος του βραβείου Ζαχάροφ να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική. Με αυτό το θέμα, στην ουσία, θίγουμε και πολλά άλλα πολύ σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, με τη διεθνή συνεργασία σε περιοχές συγκρούσεων. Δεν είναι μόνο το θέμα των μετάλλων αυτών που αναφέρει το κείμενο, αλλά και πολλά άλλα. Στην επόμενη ολομέλεια θα μιλήσουμε για τα κλωστοεφαντουργικά στον Μπαγκλαντές. Τι θέλω να πω. Πρέπει να εξετάσουμε τα διάφορα θέματα της εμπορικής μας πολιτικής και να επιδείξουμε μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ τους. Ο προηγούμενος επίτροπος Ντεχνίχτε όταν επισκέφθηκε τον Μπαγκλαντές είπε πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα μέτρα. Το επιτύχαμε εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αυστηρότεροι και γι' αυτό κάνω έκκληση και ελπίζω μέσω της περαιτέρω συνεργασίας για το θέμα αυτό να καταλήξουμε σε μια υποχρεωτική εφαρμογή. Και αυτό έχει να κάνει και με τον νόμο Dodd-Frank. Ο κύριος Βίνκλερ είπε ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των επιπτώσεών του ανάλογα με την ε, άποψη του κανός και την, ε, τις πηγές πληροφόρησης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Ποια ήταν αρχικά η πρόθεση τι ήταν δυνατό μετά από ένα χρόνο, όλα αυτά να τα εξετάσουμε. Υπάρχει, υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ε, δρούν οι αμερικανικές εταιρείες σε αυτήν την περιοχή, ούτως ώστε να μην συμβάλλουν στην επιδείνωση. Και βεβαίως είμαι υπέρ μιας παγκόσμιας αλυσίδας ε, διανομής των προϊόντων. Αυτό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έμα, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τι εννοώ. Ακριβώς επειδή πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες, γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε συνολικά και παγκόσμια με την αλυσίδα διανομής αυτών των προϊόντων. Πρέπει να καθορίσουμε σαφώς ότι πρέπει να αφορά το κείμενό μας όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και ιδίως με αυτούς που για πρώτη φορά θέτουν σε κυκλοφορία αυτά τα αγαθά. Είναι ούτως άλλως πάρα πολλοί αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα ούτως ώστε να ε, συμμετέχουν και αυτοί στο σύστημα πληροφόρησης του ΩΣΑ. Αυτό θα διευκολύνει την κατάσταση. Και όλοι οι φόβοι ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς. Όχι, οι καθευτήρες γραμμές τους επιτρέπουν ε, να εξηγήσουν ότι δεν μπορούν άμεσα να προσαρμοστούν και να δίνουν τις πληροφορίες αυτές όλες Υπάρχει ένα διετές, ε, υπάρχει μια διετής περίοδος προσαρμογής. Επίσης, επειδή υπάρχουν οι φόβοι του συναδέλφου Βίνκλερ σε σχέση με τον νόμο Dodd Frank, είπαμε Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε ποιε είναι οι περιοχέ ε, συγκρούσεων και μετά θα αναλάβει τι ευθύνε τη Κομισιόν. Αυτά λοιπόν και παραλαμβάνω από πλευρά μα. Θέλουμε να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα με βάση αυτά που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Thanks a Ευχαριστώ, λέει κυρία Κέλλα. Πολύ καλή συνεργασία μας με τον εισηγητή. Η πολιτική μας ομάδα θέλει να καλύψει όλη την ε, αλυσίδα, να είναι υποχρεωτική η ρύθμιση, να μην επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα. Πάντως εμείς θεωρούμε ότι για να πετύχουμε το στόχο μας κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Συμφωνούμε με αυτό και θα το πετύχουμε μόνο εάν γίνει υποχρεωτική ρύθμιση για όλη την αλυσίδα. Και έτσι να λάβουμε υπόψη για τις ΜΜΕ. Είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε και όσον αφορά την προσφορά τα βασικά σημεία τις εξορίξεις, τα δηληστήρια και αυτά όλα επισημάνθηκαν και αναφέρθηκαν προηγουμένως ότι δηλαδή θα πρέπει δε να προσέξουμε όχι μόνο την κορυφή της της παραγωγικής πυραμίδας, της προσφοράς μάλλον, της πυραμίδας, αλλά θα πρέπει όλη την αλυσίδα να την καλύψουμε. Η ιδέα λογική του να καλύψουμε όλη την αλυσίδα και όλες τις εταιρείε ότι να χρησιμοποιήσουν όλες οι αλυσίδες, όλες οι τρεις αλυσίδες, την μόχλευση και να μπορέσουν να προσχωρήσουν στην δέουσα επιμέλεια. Και επίσης να εξασφαλίσουμε το ότι η σχέση αυτή που υπάρχει τώρα θα αλλάξει. Και αυτό είναι ο στόχος των όσων προσπαθούμε να πετύχουμε. Επίσης πάλι για το κριτήριο της ε, δέουσας επιμέλειας, αν δείτε τις καθηγητές γραμμές του ΩΣΑ, θα διαπιστώσετε ότι προβλέπονται αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν με αρκετή ευελιξία και οι εταιρείε θα πρέπει πρώτα πρώτα να επισημάνουν στην προσφορά ποια είναι, ποιες είναι αυτές οι εγκαταστάσεις των ε, ε, μεταλλουργίων αυτών και επίσης να μην ξεχνούμε ότι οι εταιρείε δεν θα υποστούν κυρώσεις αν αμέσως δεν μπορέσουν να δώσουν τις ε, σχετικές πληροφορίες. προ... Ε, δέουσα επιμέλεια αυτό σημαίνει. Προοδευτική εφαρμογή. Βαθμία. Έτσι θα γίνει το πράγμα. Τώρα. Να μην τα παραλάβω, αλλά μόνο εάν καλύψουμε όλη την αλυσίδα δεν θα έχουμε τις ε, στρεβλώσεις. Αλλιώς θα υπάρχουν κίνητρα εισαγωγής πρώτων υλών. Και θα έχουμε 240 μεταλλουργία εκτός. Όσον αφορά το ότι θα στραφούν αυτοί στην Ασία και όχι στην Ευρώπη. Για την ΜΜΕ να επαναλάβω τα ίδια. Τώρα για να δούμε τι γίνεται με άλλους φυσικούς πόρου θα πρέπει να καλύψουμε. Ναι, λέμε και εμείς Γιατί η χρηματοδότηση των συγκρούσεων δεν περιορίζεται μόνο εδώ. Παντού γίνεται αυτό. Και αφορά την πρόσβαση και αφορά όλους τους φυσικούς πόρους. Άρα να τους καλύψουμε όλους. Θα πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες ήταν οι συνέπειες του νόμου Dodd Frank. Είχε πεδίο εφαρμογή γεωγραφικά περιορισμένο. Γι' αυτό και μετακινήθηκαν οι εταιρείε. Άρα εμείς τώρα θα πρέπει να καλύψουμε πολύ περισσότερη περιοχή. Ναι, θα τα φορτώνουμε όλα στο όνομα του Τούτφρεν. Επίσης υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα γύρω στο τι ισχύει. Δεν ξέρω οι τι ισχύει. Άρα αυτά τα λάθη μην τα επαναλάβουν. Ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, εισηγητή Συνάδελφοι, για να πετύχουμε λοιπόν το καλύτερο αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της βίας, ε, υποστηρίζουμε αυτή την διάταξη για την τέουσα επιμέλεια. Αλλά πολύ λυπάμαι που δεν έγινε πλήρως κατανοητή η πρότασή μας. Για παράδειγμα, σαν αφορά τα συνδικάτα. Για να εξηγήσουμε πώς το σύστημα των Frank επηρεάζει τις Ιταλικές εταιρείε. Η πρότασή μα δεν είναι ένα ευρωπαϊκό νόμο, Ρόδο Φρανκ. Είναι ένα διαφορετικό τελείω σύστημα. Άρα, καλύτερα θα ήταν να δώσουμε μία επισκόπηση δομαστικών στοιχείων. Καταρχά, προτείνουμε υποχρεωτικό κανονισμό. για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, όπω έχει φανεί τώρα, δεν θα κάνω καταβάλει επαρκή προσπάθεια παρά τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπάρχουν. Εκτός και αν υπάρχει νομική απέτηση. Το βασικό θέμα επίσης έχει να κάνει με τη συμμετοχή όλων των φορέων για να υπάρχει δέουσα επιμέλεια σε όλη την αλυσίδα παραγωγής από την πηγή μέχρι τον τελικό προορισμό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καλύπτεται από όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή θεωρεί ότι οι εισαγωγή είναι ε, εισαγωγή συμμετέχουν στη διαδικασία ανεξάρτητα από την διαδικασία και την αλυσίδα παραγωγή. Στην πρότασή μα, λοιπόν, Αντιθέτω. ε, αναφερόμαστε μόνο στα μεταλλουργία Ω φορεί. Και θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα σημεία τα κρίσιμα με την μικρότερη γραφειοκρατική προσπάθεια. Άρα το μοναδικό επιπλέον καθήκον για μια μικρή επιχείρηση που πουλάει σε χρυσό για παράδειγμα θα είναι ένα τηλεφώνημα στον άμεσο προμηθευτή του για να βεβαιωθεί ότι ο προηγούμενο του στην αλυσίδα παραγωγή ε, και πιάνει ταυτότητά του. Ζητώντα το όνομα του μεταλλουργίου, για παράδειγμα, ή τη εγκατάσταση τήξη, τη εγκατάσταση ε, εξευγενισμού. Αυτό είναι μια μικρή προσπάθεια για τις μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή εδώ στην Επιτροπή μας. Ή θα επιλέξουμε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου υπάρχει ένα θελούσιο σύστημα το οποίο εκφίσως δεν είναι ε, υποχρεωτικό αλλά είναι και κοστοβόρο εφόσον αποφασίσουν να το εφαρμόσουν ή θα υποστηρίξουμε ένα σύστημα υποχρεωτικό για όλου του φορεί, αλλά εύκολο, που δεν θα επιβαρύνει κάποιου πιο πολύ από ό,τι άλλου, ιδιαίτερω ε, τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ε, στη μία περίπτωση θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα εφαρμόζεται από όσου ε, ήδη εφαρμόζονται δέουσα επιμέλεια τι μεγάλε επιχειρήσει, αφήνοντα κατά μέρο τι μικρέ επιχειρήσει και αφαιρώντα του δυνατότητα συμμετοχή σε δημόσιε συμβάσει, Από την άλλη έχουμε ένα σύστημα συνολικό ε, εύκολο και το οποίο απευθύνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν το έλαβε καν υπόψη αυτό ως ε, λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ φοβάμαι ότι υποστηρίζει κάποια περιορισμένα συμφέροντα επειδή αυτό λειτουργεί ο σύστημα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, δεν θα κανεί άλλο το λόγο. Και ω εκ τούτου θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Χαράτσο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλιά τους. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον ε, με το οποίο ασχολείται το Κοινοβούλιο. Έχουμε ηθική υποχρέωση να ασχολούμεθα με την παραγωγή αγαθών από αυτές τις περιοχές συγκρούσεων και να μάθουμε και από τα λάθη του παρελθόντος και να έχουμε μια λειτουργική λύση αλλά και αμερόληπτη. Το είπε και ο κύριος Βίνκλερ. Να βρούμε τα σωστά μέτρα τώρα για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους είναι δύσκολο καθήκον. Εξετάσαμε πολλές από τις επιλογές που και εσείς εξετάζετε σήμερα κατά την ε, εκπόνηση της πρότασης. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τις προτάσεις σας και εργαζόμεθα για να δούμε πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις προτάσεις σας στα συνοδευτικά μέτρα. Χθες πήρατε σαφή δέσμευση από, τον αντιπρόεδρο, από την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη και τους Επιτρόπους Βάλτσον και Νίμιτσα ότι θα δώσουμε οικονομική βοήθεια για την υπεύθυνη εξόριξη σε αυτές τις περιοχές και κατεργασία. Θα πολλαπλασιαστεί επί πέντε η βοήθεια που δίδεται για τους στόχους αυτούς. Να αναφερθώ σε μερικά σημεία και σε μερικές ερωτήσεις που θέσατε. Γιατί η Επιτροπή δεν προτείνει υποχρεωτικό σύστημα για τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει στρέβλωση του εμπορίου και μείωση της δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές συγκρούσεων. Μπορεί να είναι αυτό και ένα μειονέκτημα στον ανταγωνισμό για τα περαιτέρω στάδια της κατεργασίας και εμπορίου. Και να μην έχουμε και προβλήματα ε, ασφάλειας προμήθειας, ασφάλειας εφοδιασμού για τις χώρες μας. Αυτή η κίνδυνοι χωρίς ε, προπαρασκευαστικές, προκατακτικές ε, μελέτες αντικτύπου είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε τι θα γίνει και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σόφρονες. Και σόφρονες σημαίνει εθελοντικό σύστημα και επίσης κίνητρα για να συμμετάσχουν περισσότερες στο σύστημα. Τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε οι εταιρείε που θα συμμετάσχουν σε αυτό το εθελούσιο σύστημα θα κάνουν υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών. Πρώτα απ' όλα υπάρχει δημόσιο αίτημα για τέτοια υπεύθυνη ε, προμήθεια. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία δίνοντας νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο συνδεδεμένο με ένα πακέτο κινήτρων τα κίνητρα αυτά είναι τμήμα του πακέτου. Θα είναι για παράδειγμα να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες ε, μέσω διπλωματικών και αναπτυξιακών ε, κινήτρων. Άμα ακούσετε τους εκπροσώπους του κλάδου, τους οποίους νομίζω έχετε συναντήσει επανειλημμένα, έχουν συνέστηση του πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα κίνητρα, να βοηθήσουν την αγορά. Επίσης εξετάζουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Για παράδειγμα, να ενισχύσουμε την μη ε, οικονομική γνωστοποίηση δραστηριότητας, ιδίως για τις μεγάλες εταιρείες, και να συμπεριλάβουμε αυτήν την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών στη σήμανση των προϊόντων μας. Ενισχύουμε όποιες προσπάθειες γίνονται επιτόπου για τέτοια προσέγγιση για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν με βάση τη δική μας προσέγγιση. Όχι μόνο στην περιοχή των μεγάλων λιμνών, αλλά και ευρύτερα. Τώρα έγιναν κάποια σχόλια σήμερα. Ιδιαίτερα τα σημεία όπου υπάρχουν συμφορήσεις. Είναι οι εγκαταστάσεις τήξης, οι εγκαταστάσεις εξεργενισμού, μετατροπής, αλλά αντίθετα από αυτά που είπε η κυρία Άγενα, δεν υπάρχει δυστυχώς φαινόμενο ντόμινο, όπως είδαμε από τη μελέτη αντικτύπου και από την εφαρμογή του νόμου Dodd Act. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία εφοδιασμού. Γι' αυτό η Ένωση με τις προτάσεις της προτείνει ένα κατάλογο των εγκαταστάσεων τήξης Παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι μόνο για τους ε, ενωσιακούς, ε, τις ενωσιακές τήξης και μετατροπής. Αυτό είναι ευρύτερο από αυτά που προτείνει ο ΣΑ. Δεν υπάρχει τέτοιος κατάλογος στα δικά τους μέτρα και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας γι' αυτό. Και κάτι άλλο που πηγαίνει παραπέρα από τις καθευτήριες γραμμές του ΩΣΑ είναι οι δομές για την ε, εφαρμογή μέσω των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Αυτό δεν το λέει ο ΩΣΑ στα μέτρα του για την δεωση επιμέλεια. Αυτό που η κυρία Μακλάρκιν για το εγχειρίδιο. Ναι, το εκπονούμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και αναλυτική ανάλυση του λογιστικού ελέγχου. Τελευταίο γιατί η υποχρεωτική προσέγγιση για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού δεν θα ήταν σκόπιμη. Πρώτα απ' όλα αυτό θα σημαίνει ότι θα συμμετείχαν ε, πολλές, ενδεχομένω εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ένωση, κυρίως μικρομεσαίες και αξιόλογο κόστος. Αυτό θα προκαλούσε διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να είχε ως επίπτωση απαγορεύσεις εισαγωγών από τις χώρες προέλευσης που δεν ήταν μόνο η ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Οπότε σας καλώ κύριοι βουλευτές να λάβετε υπόψη τα επιχειρηματά Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βίγκλερ, θα θέλατε. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι και Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συζήτηση και τις προτάσεις σας για τα όσα σχολιάζατε και χαίρομαι που ακούω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες υπεύθυνε εγκαταστάσεις γιατί στο, στο, στο, στο εγχειρίδιο που θέλουμε ε, θα, θα χαιρόμουν ακόμη περισσότερο εάν είχαν προηγηθεί αυτές, αυτά τα σχόλια, αυτές τις προσπάθειες για την, ε, ε, για την, για την λίστα των υπευθύνων βιομηχανιών ε, τώρα έχουμε τις τροπολογίες, οπότε εντάξει, να δούμε τι θα γίνει με την διαφάνεια. Η διαφάνεια βλέπουμε ότι είναι το ζήτημα εκείνο το οποίο απασχολεί τους Ευρωπαίους και για το TTIP, για τις εμπορικές εγκαταστάσεις, για την επίλυση των ε, ε, διαφορών παντού. Και γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω εκείνη την προσέγγιση αυτούς που λένε δηλαδή ότι μπορούμε να έχουμε δημιουργεί δυνατότητα στις περιοχές συγκρούσεων. Μπορείτε ότι μπορούμε εκεί να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και ότι μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν κράτη που λειτουργούν εύρυθμα με το εμπόριο και με υποχρεωτικές ρυθμίσεις που θα φορούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν το καταλαβαίνω, στο μέλλον θα προσπαθήσω να δείξω περισσότερη προσπάθεια κατανόησης, αλλά τέλος πάντων τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να συμβιβαστούμε και τελειώνοντας πρόεδρε θέλω να πω ότι αντιδρούν θετικά οι Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδων επιχειρήσεων Και όταν προβαίνουμε σε αξιολόγηση της επιχείρησης και έχουμε αυτές τις επιστολές των πυρογνωμών που μας έρχονται εδώ σε αντίδραση και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα βαρύνει για την απόφασή μας. Ο πρόεδρος. Κύριε Βίντε, ευχαριστούμε πολύ και καλή τύχη την επόμενη εβδομάδα για την έκθεσή σας. 14 Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο. 15. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Θεωρεί ότι χρειάζεται κάποιο είδου ενημέρωση για Μεξικό, Καναδά, Ινδία. Για τις Ναι, λέει ο κύριος Κάμπελ, να σας πω μια που πιέζει ο χρόνος σύντομα, διότι είχα μια σειρά συναντήσεων με τον πρέσβη της ε, Ινδίας όσον αφορά τα εμπορικά ζητήματα. Ε, με την πρώτη εποπτική ομάδα, πρώτη Μαρτίου. Πρώτη φορά μέσα σε δύο χρόνια. Και είχαμε και τον, και τον κύριο Μπεθέρο που ήταν επικεφαλή των προγραμματεύσεων και τη εξωτερική υπηρεσία ε, την προστάμε την κυρία Φερνάντες που συμμετέσχουν αυτοί και οι δύο σε αυτήν την τόσο παραγωγική συνάντηση. Πρόκειται οι Ινδοί να πάνε σε Γαλλία, Γερμανία, όχι στις Βρυξέλλε. Άρα τι θα γίνει με την συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωση Ινδία, Είναι αυτό το θέμα το οποίο εκκρεμεί. Αρκετό καιρό Πάντω υπάρχουν πολλέ δυνατότητες. Έχουμε 8% πρόβλεψη ανάπτυξη και έχουμε 200 εκατομμύρια αύξηση πληθυσμού τα επόμενα 15 χρόνια. Άρα η αγορά αυτή προσφέρει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Οπότε προβλήματα σε πέντε τομεί. Πρώτα-πρώτα στου του δασμού, τι υπηρεσίε, έχουμε 150% ε, αύξηση σε στα, στα, στα κρασιά και στα το δίποτα. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό σαν ε, έμεσος φόρος ή σαν δασμός. Οπότε θέλουμε να υπάρχει κάποια εμπορική συμφωνία, να είναι φιλόδοξη, αλλά τελικά δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε στο 0%. Όμως η μείωση αυτών των δασμών θα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτή την συμφωνία. Επίσης ε, αυτοκίνητα και χώρες στάθμευση σημαντικό και αυτό, γιατί πρέπει Σύγχρονα στα ανταλλακτικά και στα αυτοκίνητα είναι σημαντικό να πετύχουμε κάτι και θα πρέπει να υπάρξει συμπαράσταση όσον αφορά τη συμφωνία από τους αντίστοιχους κλάδους στην Ευρώπη. Υπηρεσίες, ε, λιάνο εμπόριο και εδώ προχωρούμε για να δούμε πώς θα ανέβει το 49% για τις ε, ασφάλειες όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού. Έχουμε επίσης ε, τώρα τη, το ότι μπορούν να έρθουν δύο, δύο χρόνια στην Ευρώπη, επίσης προστασία δεδομένων και επάρκεια δεδομένων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά τις ε, ε υπηρεσίες που υπηρεσίες υποστήριξη των ειδών προ τι Ευρωπαϊκέ Εταιρείε, επίσης ε, κυβερνητικές προμήθειες και διαγωνισμοί, πολύ βασικό τώρα, γιατί είχαμε κάποιους ομοσπονδιακούς νόμους κατά της ε, διαφθοράς υπήρξε υποστήριξη, αλλά αυτή η δεν αδυνησία πρέπει να ξαναθεσπιστούν, ε, πνευματική ιδιοκτησία. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σχετικό ινδικό δίκτυο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα, παρά το ότι ε, στον ΠΟΕ υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις όσον αφορά το κατά πόσο συμμόρφωνται την Ινδία. Το θέμα των γεωγραφικών ειδήσεων επίσης είναι πολύ περίπλοκο από ό,τι μου είπαν. Τέλος, όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό είναι το πιο ακαθόδες. Γιατί θέλουμε να συμμορφωθεί η Ινδία με τις σχετικές ρήτρες. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολική αυτή η απέτηση. Πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό η Ινδία. Άρα ένα θέμα που θα πρέπει να το επιλύσουμε. Αμελικά λόγια, σε αυτό σημείο βρίσκονται ε, τα πράγματα όσον αφορά την συμφωνία με την Ιδία Προωθούμε το αιτήμα των όσων είναι περισσότερο. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε στην Ιδία Τρέχει εκεί πολύ καλά η, ανάπτυξη, καλού ρυθμού και έχει και έναν πολύ, αυξημένο, πολύ μεγάλο πληθυσμό. Ε, Βεβαίω πολλέ ε, δυνατότητε, λέει ο πρόεδρο. Αλλά όπω μα τα λέτε, μάλλον σκούρα φαίνονται τα πράγματα για το εγγύ μέλλον. Και σα ευχαριστώ. Τουρκία. Εγώ έχουμε τίποτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας ε, παρουσιάσω από πλευρά του κυρίου Παρέλη τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση στις 5 ε, Μαρτίου. Ήταν η δεύτερη συνάντηση της ε, ομάδας παρακολούθησης από τη σύστασή της και Είχαμε δύο γενικού διευθυντέ από την DigiTrade και την Digineer για να μα παρουσιάσουν τι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δεύτερη συνάντηση δόθηκε ευκαιρία να ακούσουμε και την τουρκική πλευρά. Ο γενικό διευθυντή και ο εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου που είναι υπεύθυνο για τι διαπραγματεύσει από πλευρά της Τουρκία. είχε προσκληθεί και παρουσίασε την άποψη τη χώρα του για την Τελωνιακή Ένωση και τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, να σας ε, υπενθυμίσω ότι έκανε σχετική έκθεση η Παγκόσμια Τράπεζα τον προηγούμενο Απρίλιο και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια κοινή έκθεση για την ε, διαδικασία ενημέρωσης της ε, Τελωνιακή Ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Έξι μέλη ήρθαν στην συνάντηση, πολύ καλή συμμετοχή για τέτοια ομάδα παρακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο για το Εκουαδόρ. Έλμουτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Χθε είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Δεύτερη φορά κατά αυτή τη θητεία. Για το Εκουαδόρ συγκεκριμένα. για την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με την συμμετοχή της ε, συμμετοχής ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Κολομβίας και Περού για το Εκουαδόρ, α, του Εκουαδόρ. Θα έχω μια συνάντηση της Επιτροπής Εμπορίου τον Ιούνιο-Ιούλιο και μέχρι τότε ελπίζουμε να υπάρχει μια σαφής θέση των τριών χωρών συνένωση για την ε, ένταξη του Εκουαδόρ σε αυτή τη συμφωνία. Προτείνω να συντάξουμε ένα ψήφισμα το δεύτερο εξάμεινο, καλώντας αυτή η διαδικασία να προχωρήσει. Και χθε συζητήσαμε για τις εμπορικές σχέσεις με το Περού και την Κολομβία. Θα μπορούσαμε να διευρύνουμε αυτή τη συζήτηση και με το Εκουαδόρ και μετά τη συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης άκουσα ότι ο Υπουργός ε, Εμπορίου του Εκουαδόρ θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, θα επιχειρήσω να τον συναντήσω για να ενημερωθώ για τη θέση του Εκουαδόρ για το θέμα αυτό. Okay. Πρόεδρος, ωραία ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρουσίαση στα πλαίσια του σημείου 15, 16 διάφορα, δεν θέλει κανείς να βρει τίποτα. Το σημείο 17. Οι επόμενες συνεδριάσεις 13 και 14 Απριλίου. Σας εύχομαι ε, καλό Πάσχα και καλή ξεκούραση.